Καλησπέρα σας. Ας ξεκινήσουμε. Να προχωρήσουμε στις συνήθεις ανακοινώσεις καταρχάς. Η συνάντησή μας ε, περνάει κατευθείαν στο ίντερνετ. Σας το λέω γιατί είμαι υποχρεωμένος γι' αυτό. Όπερ και γέννητο. Λάβατε την ημερήσια διάταξη. Μια μικρή αλλαγή υπάρχει στο κείμενο που λάβατε. Ο κύριος Μπροκ δεν μπορεί να είναι παρόν απόψε. Άρα, η συζήτηση για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης αναβάλλεται για αύριο. Αυτό μας επιτρέπει να δουλέψουμε απόψε κάπως πιο άνετα. Ο εισηγητής για το σημείο 12 τη σημερινή διάταξη, ο κύριο Φόξ, μα είπε ότι δεν είναι σε θέση να προετοιμάσει την έκθεσή του μέχρι αύριο. Άρα, χρειάζεται να αναβάλουμε την εξέταση του θέματος σε μια άλλη συνάντηση. Ίσως την έκτακτη συνάντηση της 17ης Μαΐου στο Στρασβούργο. Αυτές είναι οι προκαταρτικές ανακοινώσεις μου. Επί της ουσίας, θα ξεκινήσουμε με κάποιες ανακοινώσεις. Κατόπιν θα συζητήσουμε την έκθεση Χαουρέγκουι για την ε, προσχώρηση στην ΕΣΔΑ. Κατόπιν την έκθεση Μάρτιν για τις αλλαγές στον κανονισμό μετά τη συνθήκη της Λισαβόνας. Θα ακούσουμε το συνάδελφο Τσβιέφκα και θα ψηφίσουμε τις τροπολογίες για την έκθεση σχετικά με την βελτίωση της νομοθεσίας και τέλος, έγκαιρα ελπίζω, θα γίνει ανταλλαγή απόψεων για την πρωτοβουλία πολιτών. Τα υπόλοιπα περνούν πάνε για αύριο. Ανακοινώσεις. Πρώτον, μπορεί να το ξέρετε, αλλά στις 24 Απριλίου απεβίωσε στην Αθήνα ο, κύριος, ο καθηγητής κ. Δημήτρης Τσάτσος, ε, ευρωβουλευτής, εξαιρετικά αγαπητός και αξιόλογος εκπρόσωπος του Κοινοβούλιο, μέλος της Επιτροπής μας από το 1994 μέχρι το 2004. Απέστειλα μια επιστολή εξ ονόματός σας, επιστολή συλληπιτήριο προς την οικογένειά του. Νομίζω ωστόσο ότι θα ήταν ε, σκόπιμο να κρατήσουμε ενός λεπτού σιγής για να τον θυμηθούμε. Ecco. Riprendiamo i lavori. Συνεχίζουμε τις εργασίες μας. Στη συνάντηση της 19ης Απριλίου η Επιτροπή μας άκουσε τον Επίτροπο κ. Σεύκοβιτς ο οποίος μας παρουσίασε το πρόγραμμα για το 2011 σχετικά με τα θεσμικά ζητήματα. Οι συντονιστές συναντήθηκαν και εξέφρασαν την άποψή τους ότι πρέπει να αποσταλεί μια επιστολή προς τη διάσκεψη των Πρόεδρων των Επιτροπών, κάνοντας μια αξιολόγηση του τρόπου παρουσίασης και του προγράμματος αυτού. Το σχέδιο επιστολής σας έχει διανεμηθεί, το έχετε στα χέρια σας. Θα έλεγα λοιπόν, αν μέχρι το βράδυ δεν λάβω παρατηρήσεις ή σχόλια που να ζητούν δυο θόσεις ή αλλαγές, θα υπογράψω την επιστολή αυτή και θα την αποστείλω στην διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών. Λάβαμε μια σειρά αποφάσεων που αφορούν, αφορούν μια σειρά θεμάτων που συζήτησαν οι συντονιστές 27 για τους εισηγητές, ιδίω σε ό,τι αφορά την πρωτοβουλία πολιτών. Η επήλθε συμφωνία με την επιφύλαξη της έγκρισης από τη διάσκεψη των Προέδρων να είναι δύο εισηγητές ειδικότερα ο κύριος Λαμασούρ και η κυρία Γκουρμάη. Η έκθεση αυτή έχει αξία τριών πόντων για τον κάθε ένα φαντάζομαι εισηγητή. Κατόπιν υπήρξε συμφωνία για το αίτημα της Επιτροπής Αναφορών να μετάσχει στις εργασίες σαν συνεργαζόμενοι με βάση το άρθρο 50 του κανονισμού Επιτροπή. το θεώρησαν σκόπιμο αυτό οι συντονιστές. Επίσης ζητήθηκε να προτείνουμε στο Κοινοβούλιο να υπάρξει διαβούλευση για το ίδιο θέμα, την Πρωτοβουλία Πολιτών δηλαδή, με την Επιτροπή Περιφερειών και την Οικονομική Κοινωνική Επιτροπή. Σε ό,τι αφορά την διοργανική συμφωνία για τη συνεργασία στα θέματα του προπολογισμού, καμία ομάδα δεν πρότεινε εισηγητή. Άρα ο υποφαινόμενος χρειάζεται να αναλάβει την γνωμοδότηση που βεβαίως δεν έχει αξία μηδέν πόντους. Σε ό,τι αφορά την ενεργοποίηση του άρθρου 291 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ένωσης, που αφορά τα εκτελεστικά μέτρα, ορίστηκε ως εισηγητής προς γνωμοδότηση ο κύριος Φόξ. Είπα προηγουμένως ότι ε, επήγει το ζήτημα της γνωμοδότηση αυτή, αλλά η αρμόδια επιτροπή, νομική, στην αρμόδια επιτροπή, την νομική επιτροπή, ο κύριος Φόξ ζήτησε την αναβολή ωστόσο και αποφασίσαμε να συζητήσουμε το θέμα στην έκτακτη συνάντηση που προβλέπεται για τη συνεδρίαση του Στρασβούργου, στην Ολομέλεια του Στρασβούργου. Σε ό,τι αφορά την αλλαγή των χρηματοοικονομικών κανονισμών και κανόνων για την υπηρεσία εξωτερική δράση και εδώ μια προφανής παρατηρήσει είναι ότι ο καταλληλότερος για τη γνωμοδότηση είναι αυτός που έχει την ευθύνη συνολικά για την ε, έκθεση για την υπηρεσία εξωτερικής δράσης και πρότειναν τον συνάδελφο κύριο Φερχόφστατ οι συντονιστές. Τελευταίο θέμα, πρέπει να ορίσουμε από το ΕΛΚ, δεν ξέρω αν το έκανε το ΕΛΚ την αίτηση αυτή, πάντως πρέπει να ορίσουμε εισηγητή για την, εφαρμογή, την έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του 51 του κανονισμού που αφορά στις ε, μικτές συνεδριάσεις επιτροπών. Η διάσκεψη των πρόεδρων επιτροπών ανέφερε στην Επιτροπή μας να εξετάσει το θέμα και να προτείνει πώς μπορεί να λυθεί το ζήτημα με καλύτερο τρόπο. Η ομάδα του ΕΛΚ ε, ζήτησε τον να αναλάβει, να, να δώσει αυτό τον εισηγητή, αλλά δεν έχουμε όνομα ακόμα. Περιμένουμε με παράκληση να μας δοθεί το όνομα να σας ενημερώσω ότι όπως συμφωνήθηκε από τους συντονιστές, για να προετοιμαστούν οι εργασίες του εισηγητού συναδέλφου κ. Ζαυκόφσκη για, την, για τις μονομερείς δηλώσεις που σε πολλές περιπτώσεις εκφράζουν και προσθέτουν τα κρατη στις αποφάσεις που λαμβάνονται συλλογικά. Ο κύριος Τρακόφσκι ζήτησε να μπορεί να χρησιμοποιήσει να οργανώσει μια μελέτη για να ξέρει τη συχνότητα και τις συνέπειες αυτών των μονομερών δηλώσεων, δηλαδή πόσες έγιναν και τι συνέπειες είχαν. Σωστό το θεωρούμε και συμφώνησαν με την πρόταση αυτή οι συντονιστές. Άρα μπορούμε να προχωρήσουμε στο πρώτο θέμα ουσίας. Συγγνώμη. Πρόεδρε, με συγχωρείτε. εισαγωγή που κάνετε περισσότερο τη σειρά των εργασιών θέτει. Και θέλω να θέσω στους συναδέλφους το εξής. Την ανάγκη να εξετάσουμε γρήγορα σχετικά το θέμα που αφορά τον ενιαίο τρόπο ψηφοφορίας σε ευρωπαϊκό πλαίσιο, που είναι αρμοδιότητα της Επιτροπής, για να αποφύγουμε να συζητήσουμε το θέμα αυτό ένα χρόνο πριν τι εκλογέ και να μην κάνουμε πάλι τίποτα. Επειδή θα χρειαστεί να υπάρξει μια διεξοδική συζήτηση για να γίνει ομοιογενής ε, ο τρόπο εκλογής, θα πρότεινα στην Προεδρία να το λάβει υπόψη και να κρίνει όταν ε, θεωρεί σκόπιμο, αλλά το συντομότερο δυνατό, την ε, κίνηση των διαδικασιών. Σωστό αίτημα. Η συνθήκη της Λισαβόνας προβλέπει ότι πρέπει να υπάρχει ενιαίος εκλογικός νόμος. Ο κανονισμός αναθέτει στη δική μας Επιτροπή την σχετική αρμοδιότητα. Στην προηγούμενη θητεία ο συνάδελφος κ. Ντάφ είχε υποβάλει ένα κείμενο που κατόπιν ε, κρίθηκε ότι λόγω των δυσκολιών που υπήρχε έπρεπε να αναβληθεί για τώρα, να μεταρρυθεί για την τωρινή θυσία, ε, θητεία, αλλά αποφασίστηκε να αναλάβει ο κύριος Ντάφ εκ νέου το θέμα και είναι στην ημερήσια διάταξη. Αύριο το πρωί μπορούμε να ξεκινήσουμε μια σχετική συζήτηση. Μακρά φαντάζομαι, θα το θυμάστε και στους συντονιστές ε, του συζητήσαμε και ο κύριος Ντάβ ζήτησε να υπάρξει παρέκκληση στο όριο που κανονικά τίθεται για τις εκθέσεις, δεν ξέρω πόσες σελίδες είναι, αλλά ζήτησε ότι είναι τόσο περίπλοκο το ζήτημα και απαιτεί μια δράση ε, παρέμβασης και πειθούς προς τα κράτη-μέλη, ε, τονίζοντας ότι οι, οι λεπτομέρειες του θέματος δεν μπορούν να ε, παρουσιαστούν μόνο σε ένα μικρό αριθμό σελίδων. Ζήτησε λοιπόν παρέκκληση να, έχει τη δυνατότητα να υπερβεί τα, τα όρια. Του το παρεχώρησα ήδη. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι καλύψαμε και αυτό το θέμα και προχωρούμε στην εξέταση τι θεσμικέ πτυχέ τη προχώρηση τη Ευρωπαϊκή Ένωση στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και Θεμελιωδών Ελευθεριών, την ΕΣΔΑ. Ήδη είχαμε μια πρώτη συζήτηση στις 17 παρελθόντο Μαρτίου. Είχαμε 61 τροπολογίε, Η συγητής είναι ο κύριος Ραμόν Χαουρέγγι Ατόντο. Έχουν υποβληθεί τροπολογίε για να επιλύσουμε τον, το πρόβλημα. Ο κύριος Χαουρέγγι, τον οποίο ευχαριστώ για την πολλή δουλειά που έκανε, πρότεινε 14 συμβιβαστικές τροπολογίες. Ο στόχος είναι να υπάρξει έγκριση του κειμένου στην Ολομέλεια στην Ολομέλεια του Μαΐου, της 18ης Μαΐου. Επειδή είναι σημαντικό το θέμα, θα παρακαλούσα τον συνάδελφο να παρουσιάσει τις, προτάσεις, τις συμβαστικές προτάσεις και κατόπιν θα ακούσουμε τις παρατηρήσεις των άλλων μελών. Συστήνω ωστόσο όλοι να είμαστε κάπως ε, όσο πιο συνοπτικοί γίνεται. Θέλετε να ψηφίσουμε χωρίς να κάνει παρουσίαση ο συνάδελφος. Να ψηφίσουμε. Βλέπω ότι ο κύριος Χωρέκη θέλει να μιλήσει. Θα μιλήσω. σύντομα, αλλά πρέπει να το κάνω. Όντως, Πρόεδρε, νομίζω ότι μπορούμε να ψηφίσουμε την έκθεση σύντομα. Η υποχρέωσή μου, ωστόσο, είναι να εξηγήσω σε όλα τα μέλη της Επιτροπής ότι μετά από τις δύο συζητήσεις που είχαμε στην Επιτροπή, την ακρόαση των εμπειρογνωμόνων και τη δουλειά που κάναμε με τις 61 τροπολογίες που υποβλήθηκαν. Υπάρχει, και αυτή είναι η σημαντικότερη δήλωση που θέλω να κάνω, υπάρχει συνένεση, εκτεταμένη, επαρκής πάντως συνένεση, ώστε το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή να περάσει στην Ολομέλεια μια σαφή, ξεκάθαρη θέση, ομόφωνη πιστεύω, του ότι το Κοινοβούλιο παροτρύνει, παρακινεί και ενθαρρύνει την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, όπως ε, θα είδατε από τις απαντήσεις που δόθηκαν στις 61 τροπολογίες που υποβάλλατε, ε, πολλές επειδή διευκρινίζουν, βελτιώνουν ή προσθέτουν κάτι στο, στο κείμενο, έγιναν δεκτές. Τούτο συμβαίνει με πολλές τροπολογίες των κυρίων Μέντες Βίγκο, της κυρίας Γιαννάκου, του κύριου Κασίνη, Προεδρού, του κύριου Νταφ, της κυρίας Μπελιέ και του κύριου Μέσερμιτ. Αυτό που προτείνω για την ψηφοφορία είναι να γίνουν δεκτές πολλές από τις τροπολογίες, σε πολλές περιπτώσεις να υποβάλλονται συμβιβαστικές τροπολογίες, 14 συνολικά που υπέβαλα, για να καλυφθούν πολλές από τις τροπολογίες που υποβλήθηκαν. Υπάρχουν κάποιες που δεν έγιναν δεκτές, διότι κατά άποψή μου είναι περιττές. Είτε διότι είναι περιττές, συγγνώμη, είτε διότι σε μερικές περιπτώσεις μπερδεύουν το κείμενο η ερμηνεία μου περιορίζει, η κατά, την ερμηνεία μου ε, περιορίζουν ή αντιβαίνουν στο πνεύμα της πορείας που θέλει να ακολουθήσει το Κοινοβούλιο. Τρεις διευκρινήσεις θέλω να κάνω πρόεδρε για τις τροπολογίες που θα ψηφίσουμε διότι είχα συζητήσεις μέχρι να πω και θα ήθελα να ενημερώσω τα μέλη της Επιτροπής ότι υπάρχουν τρεις αλλαγές που θέλω να υπογραμμίσω. Πρώτον, ως συνέπεια ε, συζητήσεων που είχα με την κυρία Γιαννάκου για την παράγραφο 1, 4, εδάφιο 4 της τροπολογίας αυτής, που αναφέρεται στη συμβιβαστική τροπολογία 5, να σας πω το εξής. Πρότεινα στην κυρία Γιαννάκου να αποφύγουμε να ψηφιστεί η τροπολογία αυτή, διότι πιστεύω ότι στο πνεύμα και στο περιεχόμενο σε, αντικατοπτρίζεται η ιδέα αυτή καλύτερη στο νέα εδάφιο της εκθέσεως. Θα μπορούσαμε μάλιστα να σκεφτούμε ότι μπορεί να υφίστατο και κάποια αντίφαση με μια τροπολογία που έχουμε δεχθεί την 39 τροπολογία του κ. Μέντες Δεβίγου που θέτει σαφώς ότι το δικαστήριο του Στρασβούργου, το ΕΔΑΔ, είναι το τελευταίο όργανο στο οποίο πηγαίνει κάποιο όταν έχουν εξαντληθεί όλες οι υφιστάμενες δικαστικές οδοί για το ίδιο θέμα και τα, το, εν λόγω, το εμπλεκόμενο, στο εμπλεκόμενο κράτος μέλος ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή συμπεριλαμβάνουμε και το ΔΕΚ. Η κυρία Γιαννάκου μου είπε ότι συμφώνησε με την ερμηνεία μου και πιστεύω ότι αν το δηλώσει και ευθέω, θα μπορούσαμε να το επιβεβαιώσουμε αυτό, ε, να αποφασίσουμε ότι δεν θα γίνει ψηφοφορία επί αυτή τη τροπολογία, άρα ούτε θα γίνει, δεν θα γίνει το ίδιο και στι τροπολογίε για τα εδάφια 4α και 4β που αναφέρονται στις τροπολογίες 15 της κυρίας Γεννάκου πάντα. Το ίδιο να πω και για μια τροπολογία που υπέβαλε ο κ. Κασίνη στην παράγραφο 2. Μιλώ για τη συμβαστική τροπολογία 6. Στην τροπολογία αυτή είχαμε μια συμβιβαστική τροπολογία που δεν θεωρούσε επαρκή ο κύριος Καζίνη και μέχρι πριν από λίγα λεπτά δεν μπορούσαμε να ολοκληρώσουμε. Εγώ θέλω να σας πω το κείμενο τη τροπολογία που συμφώνησα νομίζω με τον κύριο Κασίνη αλλά και ο ίδιος βεβαίως θα πρέπει να το αναφέρει Μιλούμε για μια τροπολογία που αναφέρεται, επαναλαμβάνω, στο εδάφιο 2 της εκθέσεως και παραπέμπει στην τροπολογία 6 τη συμβαστική. Αυτή η τροπολογία θα έχει μια τροπολογία που τη βλέπετε σε μαύρα χρώματα στο τέλος παραγράφου και θα λέει τα εξή. Θα τα διαβάσω στα ισπανικά, γιατί ισπανικά το έχω γράψει. Δεν νομίζω όμως ότι θα υπάρχει πρόβλημα στη μετάφραση. Στην τελική προ, Και σύμφωνα με τα άρθρα 4α και τη της 4 4.2 συγγνώμη και 6.3 της συνθήκης, πρέπει να τηρούνται οι παραδόσεις, οι συνταγματικές παραδόσεις και ταυτότητες των κρατών μελών. Αυτό είναι μια προσχώρηση που σημαίνει ότι η προσχώρηση στην παράγραφο 2 δεν περιλαμβάνει ενσωμάτωση νέων αρμοδιοτήτων όπως σαφώς το αναφέρει η συνθήκη. Η προσθήκη απλά υπενθυμίζει ότι η συνθήκη στο άρθρο 4, 2 και 6, 3 υπενθυμίζει ότι πρέπει να, τιμούνται, να τηρούνται οι συνταγματικές παραδόσεις και ταυτότητες των κρατών μελών. Μια τελευταία ένα τελευταίο σχόλιο. Ε, η τροπολογία των κυρίων Ντάφ και Ήλτσεφ. Η τροπολογία 30. Για την παράγραφο 5, εδάφιο 1. Οι κύριοι Ντάφ και Ήλτσεφ προτείνουν <clears throat> μια τροπολογία που θέλει να θέσει ότι ο ρόλος του δικαστή, του Ευρωπαίου δικαστή που θα ορίζεται από το Συμβούλιο της Ευρώπης στη συγκεκριμένη περίπτωση, θα ε, λειτουργεί ισότιμα με τους υπόλοιπους ε, δικαστές, ακόμα και όταν προσθέτει ε, μέρος μέρο τη είναι η ένωση στη συγκεκριμένη περίπτωση. Εμείς θεωρήσαμε ότι αυτό δεν είναι αναγκαίο, διότι είναι προφανές κατά την άποψή μα ότι όταν ο Ευρωπαίος δικαστής παρίσταται, εφαρμόζονται οι κανόνες που θεσπίζει η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τους δικαστές κάθε χώρας. Και ε, μία από τις υποχρεώσεις είναι η παρουσία τους. Όταν το ζήτημα αφορά το κράτος μέλος ή την Ένωση στη συγκεκριμένη περίπτωση. Εγώ θεώρησα ότι είναι περιττό και για να προσπαθήσω να καλύψω αυτό έχω μία τροπολογία που λέει απλώς τα εξή αντί για το κείμενο της τροπολογίας. Τελειώνει το κείμενο ισότιμα με τους λοιπούς δικαστές, σύμφωνα, προσθέτουμε με το άρθρο 27 παράγραφος 2 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης, που αναφέρεται ακριβώ το ρόλο των δίκαστων κάθε κράτους. Στις με τις τροπολογίες αυτές ολοκληρώσαμε το κείμενο πιστεύω. Μπορείτε να επαναλάβετε το τελευταίο λέει εκτός μικροφώνου ο κύριος Μπορείτε παρακαλώ να επαναλάβετε το κείμενο αυτό το οποίο έχετε κατατίσει. Βεβαίως. Λέμε στο τέλος της τροπολογίας σε βάση ισότητας με τους άλλους δικαστές. Εγώ, αυτό ήταν το αρχικό κείμενο της εκθέσεως. Η τροπολογία συμπεριλαμβανωμένη στις περιπτώσεις όπου ένας αντίδικος σε μία διαφορά είναι η ένωση. Εγώ προτείνω να βάλουμε σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 2 της ΕΣΔΑ που θεσπίζει ακριβώς το ότι ο δικαστής της χώρας που εμπλέκεται μπορεί να είναι παρόν. Ε, από πλευράς μου εγώ συμφωνώ με την συμπερίληψη της ε, αλλαγής στην συμβαστική πρόταση 5 που ανέφερε ο εισηγητής. Εγώ θεωρώ ότι η ταυτότητα είναι σημαντική. Αναφέρεται στη συνθήκη της Λισαβόνας και δείχνει το ότι δεν πρέπει να θυσιάζουμε την ιστορία μας. Εάν δεν υπάρχουν άλλοι που θέλουν να λάβουν το λόγο, μπορούμε να προχωρήσουμε. Να σας πω κύριε Πρόεδρε ότι θα ψηφίσουμε και θέλω να το πω στα μέλη της Επιτροπής. Θα ψηφίσουμε έλεγα τις εκθέσεις της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και Δημοσίων Ελευθεριών στον κατάλογο ψηφοφορίες εγώ αναφέρω τον τρόπο με τον οποίο κατά την άποψή μου πρέπει να αντιμετωπιστούν οι παράγραφοι των εκθέσεων αυτών. Θέλω να σας το εξηγήσω ωστόσο γιατί το λέω αυτό. Πρώτον, η έκθεση της Επιτροπής Δημοσίων Ελευθεριών, σύμφωνα με τον κανονισμό που εγκρίνουμε, που έχουμε, δεν μπορούμε, δεν μας επιτρέπει να ψηφίσουμε ελεύθερα αυτό που μας υπέβαλαν προηγουμένως οι Επιτροπευτοί. Άρα ε, προχωρούμε σε μια μορφή ενισχυμένη συνεργασία για την έκθεση αυτή. Αυτό που λέει η ΛΥΜΠΕ πρέπει καταρχήν να γίνει σεβαστό, διότι έχει το δικαίωμα να περάσει στην Ολομέλεια τις παραγράφους που ενδεχομένω εμείς ε, δεν εγκρίνουμε. Αυτό είναι ο λόγος για τον οποίο παρότι υπάρχει σύμπτωση, αναπόφευκτη σύμπτωση στις διάφορες παραγράφους έκανα μία πρόταση αποδοχής πλήρους σχεδόν των διαφόρων παραγράφων της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ διότι κατά την άποψή μου οι παράγραφοι αυτές με την εξαίρεση ορισμένων που είναι ζητήματα που αφορούν αποκλειστικά την ΑΦΚΟ, πρέπει να γίνουν σεβαστές. Στην Επιτροπή Εξωτερικών, ωστόσο, υπάρχουν πάρα πολλές παράγραφοι που, κατά την άποψή μας, ήδη εμπεριέχονται στην έκθεση της Επιτροπής μας. Για να μην υπάρχει λοιπόν επανάληψη, προτείνω να ψηφίσουμε unblock αν θέλετε, Πρόεδρε, των σημείων που δεν χρειάζεται να γίνουν δεκτές από την Επιτροπή μας και των άλλων που χρειάζεται. Εμείς λοιπόν προτείνουμε το συν ομού για όλα και το πλήν ομού για όλα, για να μην υπάρχουν επικαλύψεις στην τελική ψηφοφορία. Ευχαριστώ. Η κυρία Γιαννάκου. Euh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ ευχαρίστως θα αποσύρω την τροπολογία μου που ανέφερε ο κύριος Σορέγγι, οπότε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, συμφωνώ μαζί του. Ωραία, μπορούμε να προχωρήσουμε. Ο κύριος Νταφ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Με ανησυχεί ότι αν απλώς δεχθούμε την γνωμοδότηση της Επιτροπής Ελευθεριών ως έχει, θα υπάρξει επικάλυψη με θέματα τα οποία θίγουμε στη δικιά μας έκθεση και μάλιστα ε, συγκεκριμένα με τα ίδια θέματα θα εκφραζόμαστε δύο φορές. Χωρίς όμως να το εκφράζουμε ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Πράγμα το οποίο είναι μια πρωτοφανής διαδικασία η οποία θα δημιουργήσει μεγάλη σύγχυση. Όντως, εάν μπορούμε να ε, ε, επισυνάψουμε την γνωμοδότηση της Επιτροπής Ελευθεριών σαν συμπλήρωμα έχει καλώς. Διαφορετικά το να την ενσωματώσουμε θεωρώ ότι δεν είναι σωστό. Σωστά, αλλά ας ακούσουμε και τη γνώμη των άλλων συναδέλφων. Εδώ υπάρχουν δύο δυνατότητες λύσεων. Δεν λέμε τίποτα για την έκθεση επιτροπής ΛΥΜΠΕ. Σε μια τέτοια περίπτωση, ωστόσο, τότε, βάσει του κανονισμού που προβλέπει ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ των δύο επιτροπών, θα έχουμε δύο εκθέσεις στο τέλος. Ο τρόπος με τον οποίο θα αντιμετωπιστεί αυτό κατά την άποψή μου είναι να προτείνουμε την διαγραφή των παραγράφων της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ που προφανώς και προδήλως είναι κατά την άποψή μας περιττές διότι επαναλαμβάνουν κάτι που ήδη υπάρχει να σεβαστούμε ωστόσο το δικαίωμα της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ να κάνει την έκθεσή της. Κατόπιν θα περάσουμε στην Ολομέλεια το άθροισμα των δύο εκθέσεων έστω και αν σε κάποιους παραγράφους μπορεί να υπάρχουν παρόμοιες ιδέες. Εμείς θα βάλουμε τις παραγράφους της Λίμπε στην σειρά που τους αρμόζει για να υπάρχει μια λογική τάξη και συνέπεια διαδρομένη στην τελική έκθεση. Εγώ αυτό πιστεύω ότι να κάνουμε. Γιατί αν λάβουμε θέση επί της εκθέσεως ΛΥΜΠΕ, απορρίπτοντας πολλές παραγράφου, διότι η κατάποψή μας είναι ε, επανα, επαναλαμβανόμενες, αυτές έχουν, η ΛΥΜΠΕ έχει το δικαίωμα να πάει στην Ολομέλεια. Αυτές είναι οι συνέπειες του συστήματος ενισχυμένης συνεργασίας. Πιστεύω ότι πρέπει να το συζητήσουμε αυτό το ζήτημα, διότι εν τέλει δεν έχουμε σωστά διαρθωμένα κείμενα, κατά την άποψή μου. Δεν μπορώ ωστόσο να αποφύγω να τηρήσω αυτό που λέει ο κανονισμό. Το μόνο, η άλλη λύση είναι να μην ψηφίσουμε τίποτα από την έκθεση Λίμπερ, να το αφήσουμε στην άκρη σαν μια δεύτερη έκθεση. Δεν μπορούμε να εμποδίσουμε ωστόσο την Λίμπερ να κάνει την έκθεσή τη. Αν κατάλαβα καλά, σύμφωνα με την πρόταση του εισηγητή έχουμε δύο δυνατότητες. Ή λέμε θα υπάρχει μία έκθεση με οργανική ενότητα, άρα στην περίπτωση αυτή η τα σημεία της γνωμοδότησης της ΔΥΠΕ που είναι επί της ουσίας παρόμοια με την δική μας δεν πρέπει να ε, ψηφιστούν και να απορριφθούν με την αιτιολόγηση ότι ε, δεν ταυτίζουν, δεν έχουν ε, νόημα ή Δεχόμαστε το σύνολο της έκθεσης. Σε μια τέτοια περίπτωση θα προτείνουμε, θα μας πει ο συνάδελφος ποια είναι τα σημεία αυτά που ε, περιέχονται. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να καταψηφίσουμε την γνωμοδότη, τα σημεία αυτά της ΛΥΜΠΕ, όχι γιατί είναι αντίθετα, αλλά γιατί είναι περιτά. Η δεύτερη υπόθεση Η δεύτερη λύση είναι να ψηφίσουμε ενιαία όλη την έκθεση της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ, δεχόμενη την, την γνωμοδότηση, χωρίς να την ενσωματίσουμε τόσο οργανικά μέσα στο κείμενο. Δεν ξέρω, υπάρχουν κάποιοι συνάδελφοι που έχουν θέση επ' αυτού. Εγώ προσωπικά αλλά αυτό ο καθένα ό,τι θέλει μπορεί να πει. Θα προτιμούσε την πρώτη επιλογή. Να υπάρχει δηλαδή μία ε, ορθολογική έκθεση που δέχεται βεβαίως το περιεχόμενο της ΛΥΜΠΕ, διαγράφει ωστόσο τα σημεία που θα αποτελούν επανάληψη. Αλλά κύριε συνάδελφε, σε μια τέτοια περίπτωση πρέπει να μα λέτε Για τη γνωμοδότηση της ΑΦΕΤ πάντως δεν έχουμε προβλήματα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Τροπολογία 14. Παράγραφος 1, πρώτο εδάφιο. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία 3 του εισηγητού. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Ομόφωνα. Άρα. Καλύπτεται η 17. απέσυρε εγώ την 16. Το συμβιβαστική 4. Για το τρίτο εδάφιο της 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτό. Προχωρούμε τώρα στην τροπολογία 18, διότι 15-16 έχουν καλυφθεί, η 16 έχει, 17 ε, έχει, η 16 έχει απορριφθεί, 18 τροπολογία υπέρ, κατά, αποχές, ομόφωνα, δεκτό. Τροπολογία 19 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Προχωρούμε. Συμβιβαστική τροπολογία 5 του εισηγητού. Τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 1. Υπέρ, κατά, αποχές, μία αποχή. Κατά είστε, Ένας κατά, μία αποχή. Ευχαριστώ. Προχωρούμε. Η 15 καλύπτεται. Όλες οι τροπολογίες καλύπτονται. Τροπολογία 20 tutti i 15 sono coperti o ritirati, quindi niente. Andiamo all'emendamento. Τροπολογία 20, παράγραφος 2. Υπέρ. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική τροπολογία 6 η οποία, στην οποία έχουμε προσθέσει και την προσ, προφορική τροπολογία του εισηγητού μετά από αίτημα του Πρόεδρου. Ψηφίζουμε. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται ομόφωνα. Η 22 καλύπτεται. Και η 21 έχει καταπέσει. Ήδη καλύφθηκε από τη συμβαστική τροπολογία. 23 του εισηγητού. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δέκτη. Είκοσι τέσσερα. Εδώ έχει ζητηθεί να προχωρήσουμε σε κατά τμήματα ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα. Ποιοι είναι υπέρ του πρώτου τμήματος. Κατά. Ένας κατά. Αποχές. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται το δεύτερο τμήμα. της τροπολογίες 24 στην παράγραφο 3. Συμβιβαστική 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Μία ψήφος κατά εγκρίνεται. Τροπολογία 30. Οι άλλες έχουν καλυφθεί. Δαφ. Παράγραφος 5, πρώτο εδάφιο. Υπέρ. Α, υπάρχει μια προφορική τροπολογία. Αναφέρθηκε. Δεν χρειάζεται να το επαναλάβουμε. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 29 του εισηγητού. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Τρει ψήφοι κατά. Δεν έχουμε ψηφίσει την τροπολογία τη συμβαστική 8. Ψηφίζουμε. Ποιοι είναι υπέρ τη συμβαστική 8. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 32 καταπίπτει λοιπόν ο, ο και το 31. 33. Υπέρ της τροπολογίας 33. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 34 έχει καταπέσει. Συμβιβαστική τροπολογία 9. Στην παράγραφο 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Κανείς. Εγκρίνεται. Άρα οι 35-36 καταπίπτουν. Συμβιβαστική 10. Παρακαλώ. Μια η πολωνική εκδοχή του κειμένου είναι τελείως άσχετη. Δε, στα πολωνικά δεν έχει νόημα. Θα σας πω στα πολωνικά πως πρέπει να, να τα αναφέρουν αργότερα. Πάντως το κείμενο στα πολωνικά είναι χάλια. Αν είναι μόνο μεταφραστικό το πρόβλημα, το καταγράφουμε. Δεν αλλάζει επί της ουσίας τις άλλες γλώσσες. Ψηφίζουμε. Τη συμβαστική 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Οι 37 και οι 38 έχουν καταπέσει. 39 39 μέντες βίγκο υπέρ. Κατά. Αποχές Εγκρίνεται. 43. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται η του 43. Συμβιβασική τροπολογία 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ένα κατά. Άρα προχωρούμε στην τροπολογία 45 λέει ο πρόεδρος.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 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ε, η 42 φεύγει, το τροπολογία 46. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 47. Υπέρ, κατά, να μετρήσουμε. Επαναλαμβάνουμε την ψηφοφορία υπέρ της 47 παρακαλώ. Κατά. Εγκρίνεται. 49 τροπολογία. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 48. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβασική τροπολογία 13 του εισηγητή. Μήπως μπορεί να εξηγήσει ο εισηγητής ποιες αλλαγές προτείνει σχετικά με την αίτηση στα αγγλικά applications. νομίζω ότι ο σωστό όρο στα γαλλικά είναι ρεκέτ καλύτερα και όχι demand. Ίσως το πρόβλημα σημειώνεται σε ορισμένε μόνο γλώσσε, σε ορισμένα μόνο κείμενα. Αλλά βέβαια θα πρέπει να είμαστε όσο ακριβέστεροι μπορούμε στη διατύπωση. Ο εισηγητής για ποια τροπολογία μιλάτε ακριβώς. Στη 13 συμβιβαστική μιλάμε. Κοιτάξτε στην τροπολογία αυτή επιφέραμε διάφορες διορθώσεις. Ποια είναι αυτή που ανησυχεί τον κύριο Νταφ. Πού εμφανίζεται αυτό το κείμενο, με αυτός ο όρος που σας ανησυχεί. Ο κύριος Νταφ. Στα αγγλικά. applications. ατομικών ετοιμάτων στα ελληνικά. Και είναι η διαφορά μεταξύ προσφυγών και ετοιμάτων. Το ισπανικό κείμενο λέει petición. Εγώ δεν έχω πρόβλημα με την χρήση του όρου στα γαλλικά, demand, requête, δεν ξέρω ποιος είναι ο όρος στα αγγλικά. Εγώ δέχομαι την γλωσσική εκδοχή στα αγγλικά που προτείνει ο κύριος Νταφ. Δεν έχω πρόβλημα. Νομίζω ότι είναι ένα γλωσσικό ζήτημα. Οι λέξεις, οι όροι μάλλον έχουν το ίδιο νόημα. Ψηφίζουμε τώρα τη 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Οι 52 καλύπτονται 53. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 54, 12α, υπέρ. Κατά. Ένας κατά, εγκρίνεται. 55, υπέρ. Κατά. Αποχές, απορρίπτεται. Το 56 δεν το ψηφίζουμε γιατί είναι ίδιο με το 55. Συμβαστική 14. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Μία ψήφος κατά. Το απολογία 57. Διορθώνει ο πρόεδρος. Καλύπτεται η 57. 59. Τροπολογία. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Η μόνιμη και αξιοθαύμαστη μάχη, μοναχική μάχη του συναδέλφου κύριου Μέτερ Σμιτ. Τροπολογία 60. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 61. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 1. Για το σκεπτικό 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 3. Για την αιτιολογική σκέψη α. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Οι δύο υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Οι πέντε υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τέσσερα υπέρ κατά Με συγκινήσατε πρόεδρε και ήθελα να δείξω ελεγγύη στο συνάδελφο μέσα Σμιτ. Ε, δημοκρατία το λένε. δεν είναι δύσκολο το θάρρο αυτό. Απορρίπτεται. Τροπολογία 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 7. Μπελία. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία 1 του εισηγητού. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία συμβαστική 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τα υπόλοιπα καλύπτονται. 12 του εισηγητού υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 13. Σεβερίν υπέρ κατά εν τρεις κατά αποχές εγκρίνονται. Φτάνουμε τώρα στις γνωμοδοτήσεις των επιτροπών. Κύριε συνάδελφοι, εισηγητά, πείτε μας για την Επιτροπή Δημοσίων Ελευθεριών. Πρόεδρε, εγώ προτείνω η Επιτροπή μας να εγκρίνει όλες τις παραγράφους της ΛΥΜΠΕ με την των παραγράφων 1, 2 και 9. Η μία και οι δύο είναι ακριβώς οι ίδιες, ενώ η 9 είναι αρμοδιότητα αποκλειστική της ΑΦΚΟ και όχι της ΛΥΜΠΕ. Όλα τα άλλα, ενώ θα μπορούσαν να είναι επαναληπτικά, μπορούμε να τα εγκρίνουμε. Λάθος είναι το 7. Το 7 το υπερψηφίζουμε. Κακό στέθηκε το πλήν εδώ. Προτείνω να ψηφίσουμε σε δύο ομάδες, αν συμφωνεί η Επιτροπή μας, όλες τις παραγράφους με την εξαίρεση των παραγράφων 1, 2 και 9. Αυτό νομίζω ότι είναι αρκετό. Υπάρχει κάποιος που αντιτίθεται στην ψηφοφορία ομού. Ψηφίζουμε ομού τις τοπολογίες 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ναι, και 15. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ένας κατά δύο αποχές. Στις τροπολογίες που δεν έχουμε ψηφίσει φαντάζομαι τις, ψηφίζουμε, κατα... τις καταψηφίζουμε. Ομού επλήσεις. Ένα, δύο και 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. Τροπολογίες της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων. Και εδώ Μπορεί ο συνάδελφος ηγητή να μας προτείνει δύο ομάδε βεβαίω. Να πω στην Επιτροπή ότι ο λόγος για τον οποίο υπάρχουν περισσότερα πλήν είναι διότι στο θέμα αυτό δεν είμαστε υποχρεωμένοι να τηρήσουμε τη ε, διαδικασία του άρθρου 50. Η Επιτροπή ΑΦΕΤ δεν είναι ενισχυμένη συνεργασία, γνωμοδότηση κάνει. πολλές από τις παράγραφοι της γνωμοδοτήσεως αυτής δεν είναι ακριβώς θέμα διεθνών σχέσεων ή υπόφορουν την, προσε... προσχώρηση. Άλλες είναι. Εγώ λέω να ψηφίσουμε τις παραγράφους 2, 5, 9, 14, 15, 16 και 17 και να απορρίψουμε τις υπόλοιπες τοπολογίες. Συνάδελφοι που θέλουν να σχολιάσουν κάτι. Οι συνάδελφοι έχουν κάποιο σχόλιο. Ωραία. Ψηφίζουμε ένα πρώτο μπλοκ των τροπολογιών της Επιτροπής ΑΦΕΤ που είναι οι 2, οι 5, οι 9, οι 14, 15, 16 και 17. Υπέρ κατά, αποχές, μία ψήφος κατά και μία αποχή. Ψηφίζουμε τις λοιπές τροπολογίες. Την 3, την 4, την 6, την 7, την 8, τη 10, 11, 12, 13 αυτά. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, Απορρίπτονται. Προχωρούμε τώρα. Τελική ψηφοφορία για την πρόταση ψηφίσματος όπως τροποποιήθηκε. Υπέρ. Δεκαοκτώ. Κατά. Αποχές. 17, 18 υπέρ, ένας κατά, καμία αποχή. Συγχαρητήρια κύριε Χαουρέγγι. Και δεν είναι τυπικά τα συγχαρητήρια, κάνετε πολλή δουλειά πραγματικά. Πάντα βρίσκατε αρμονικές λύσεις σε σχέση με την θέση που ανέκυψε στην Επιτροπή σε ένα θέμα εξαιρετικής σημασίας και σπουδαιότητας. Προχωρούμε. Allora, eh, la storia di questo adeguamento e del regolamento... Η ιστορία της προσαρμογής μας στη Συνδίκη της Λισαβόνας είναι γνωστή πλέον. Ιστορικό κομμάτι είχε εγκριθεί στην προηγούμενη θητεία, πέρασε στην Ορμέλεια, εγκρίθηκε κατά το ίμιση, αναπέμφθηκε στην Επιτροπή, όπου εμφανίστηκαν αντιρρήσεις, από ό,τι φαίνεται ωστόσο ο κύριος Μάρτιν κατόρθωσε με μεγάλη ικανότητα και αυτός να βρει λύσεις που θα καταστήσουν, ελπίζω, όριμη την στιγμή για την ψηφοφορία, για την ψήφιση του κειμένου. Θέλετε να πείτε κάτι κύριε Μάρτιν ή να ψηφίσουμε. Possiamo votare. Bene. Allora. Procediamo ai voti. Devo avere... La lista di voti. Eh sì, vabbè. Allora, procediamo al voto. e λοιπόν στην ψηφοφορία. της τροπολογίας 5 που πρόκειται να ψηφιστεί σε δύο ε, τμήματα. Το πρώτο τμήμα είναι μια προφορική τροπολογία που προτείνει ο εισηγητής. Το βλέπετε, άρα δεν χρειάζεται να το επαναλάβω. Όποιος είναι υπέρ, παρακαλώ να σηκώσει το χέρι του. Ψηφίζουμε το πρώτο μέρος της τροπολογίας 5 στο άρθρο 8. δεν υπάρχει πρώτο μέρος, ε, σχολιάζει η ομίγυρης. Με συγχωρείτε, λάθος διάβασα. Πρόκειται για μία προφορική τροπολογία και ε, υποκαθιστά μία άλλη τροπολογία. Πρόκειται λοιπόν για μία προφορική τροπολογία ατού εισηγητή. Ποιος είναι υπέρ. οκτώκατα, κατά. Οκτώ υπέρ, οκτώ κατά, άρα απορρίπτεται. Θέλετε να ξαναδοκιμάσουμε. Λοιπόν, προφορική τροπολογία 5. Ποιος είναι υπέρ. 10 κατά και νέα υπέρ, άρα αυτό απέδειξε η επαλήθευση. Λοιπόν, τώρα ψηφίζουμε την προφορική τροπολογία του συναδέλφου Νταφ. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 11 στο άρθρο 37 bis. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 7 Άρθρο 74 ε, μπις. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 8. Στο άρθρο 74 τερ. Ε, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία David Μάτιν και Ρομπέρτο Gualtieri. Τροπολογία 12 ε, στο άρθρο 96 υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Τροπολογία 10. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 1, άρθρο 116 υπέρ. Κατά. Απροβάζω. Εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία Λοιπόν, μια στιγμή κύριε Πρόεδρε, στο άρθρο 117 νομίζω ότι εδώ τίθεται ένα σημαντικό θέμα. Όταν στην ε, συνταγματική συνέλευση αποφασίσαμε να υπάρξει ένα προηγούμενο, θυμάστε τι συζήτηση έγινε. Και το πετύχαμε, γιατί θέλαμε ο να υπάρχει ένας πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και τίποτα λιγότερο, δηλαδή ούτε λίγο παραπάνω ούτε λίγο παρακάτω. Αυτό που φοβάμαι είναι ότι εάν αυτός ο πρόεδρος, αν έχουμε δικαίωμα να του υποβάλουμε γραπτές ερωτήσεις και, ε, δεν, ε, ε, και δεν μπορεί να μας απαντήσει, θα είναι κάτι ακόμη παραπάνω. Και γι' αυτό πιστεύω ότι δεν είναι σωστό. Πιστεύω ότι οι συνάδελφοι διαφωνούν με την άποψή μου, αλλά σας παρακαλώ να το σκεφτείτε, διότι δεν νομίζω ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να, θέσουμε ε, γραπτές ερωτήσεις προς απάντηση από τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο κύριος Μάρτιν. Δεν θέλω να γίνει μία συζήτηση σε αυτό το σημείο. Αντιλαμβάνομαι το σχόλιο του κυρίου Μέντενς και γι' αυτό αναφερθήκαμε στις ε, γραπτές ερωτήσεις προς τον Πρόεδρο διότι ε, θα είναι για θέματα διαδικαστικά και όχι πολιτικής ενώ στα, σε προφορικές ερωτήσεις μπορούσε κανείς να τον εμπλέξει σε διάφορα θέματα αλλά σε μία ε, γραπτή ερώτηση μπορούμε να, πω, να, να λεχθεί ότι αυτό δεν είναι θέμα του Προέδρου και νομίζω ότι σαν Κοινοβούλιο έπρεπε να έχουμε αυτό το δικαίωμα να λειτουργήσουμε κατά αυτόν τον τρόπο. Ο κύριος Νταφ. Βεβαίως, μπορούμε να του θέσουμε και προφορικές ερωτήσεις διότι έρχεται στην Ολομέλεια. Δεν χρειάζεται να μας απαντήσει, αλλά εμείς μπορούμε να κάνουμε τις ερωτήσεις μας. Άρα θα πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα να συμπληρώσουμε τις προφορικές ερωτήσεις με γραπτές. Και πιστεύω ότι αν θυμάμαι τη συζήτηση η οποία έγινε ε, κατά ε, την επινόηση αυτού του ατόμου στη συνταγματική συνέλευση. Θυμάμαι πολύ καλά τι είχε γίνει και στη συνταγματική συνέλευση. Και στη συνέχεια όπως απέδειξαν τα γεγονότα, ε, διαπιστώσαμε τι ήταν το άτομο το οποίο είχαμε δημιουργήσει. Εάν λοιπόν ε, καταρτιστεί μία διαδικασία για να του θέτουμε ερωτήσεις, υπάρχει ο κίνδυνος να δώσουμε το δικαίωμα να αυξηθεί ε, το έλλειμμα δημοκρατίας. Γι' αυτό και είμαι υπέρ της επιφυλακτικής προτάσεως του εισηγητή επί του θέματος αυτού. Μέντες Δεβίγκο. Όταν έφυγε ο Φρανκ Σινάτρα, αποφάσισε να επανέλθει και ξεκίνησε με ένα, ταξί, με ένα τραγούδι λέγοντας «Ας ξαναπροσπαθήσω, let me try again». Οπότε ε, δεν υπάρχει δημοκρατικό έλλειμμα διότι έχετε τη δυνατότητα να συντάξετε γραπτές και προφορικές ερωτήσεις προς το Συμβούλιο και ε, ε, αυτοί καταρτίζουν την πολιτική ενώ ο πρόεδρος δεν είναι υπεύθυνο για την πολιτική συντονίζει, ε, ηγείται και έρχεται εδώ μετά από κάθε Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενώ πιστεύω ότι διαφορετικά θα δημιουργήσετε ένα νέο πολιτικό πρόσωπο. Το επιθυμείτε πραγματικά. Πρέπει να σας πω ότι έχετε δυνατότητα σύμφωνα με τις αρμοδιότητες του να μας εκπροσωπήσει στα θέματα της CFSP. Είναι κάτι το οποίο ακόμη δεν έχει κάνει, ενδεχομένως διότι θεωρεί ότι είναι προβληματικό. Αλλά ε, ε, είναι ε, ένας ισχυρός πρόεδρος του Συμβουλίου και όχι απλούστατα ένας, διοικητη, ένας πρόεδρος διοικητικού συμβουλίου όπως ε, καταρχήν είχε επινοηθεί. Με συγχωρείτε. Εφόσον δεν ε, υπάρχουν άλλα σχόλια μπορούμε να ψηφίσουμε. Καταρχήν την ε, προφορική τροπολογία του Ινίγκο Μέντες Vigo χωρίς την αναφορά στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Και μετά θα ψηφίσουμε και τους όρους ε, The President of the European Council που είναι η προφορική τροπολογία που προτείνει ο συγητής. Συμφωνείτε? Λοιπόν, Καταρχήν ψηφίζουμε την προφορική ε, πρόταση του Μέντες Vigo χωρίς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Άρα απορρίπτεται. Τώρα πρέπει να ψηφίσουμε την άλλη ολόκληρη προφορική τροπολογία. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Έντεκα υπέρ, δέκα κατά. Άρα εγκρίνεται. Τώρα ε, περνάμε στην τροπολογία 4, η οποία έχει ζητηθεί να ψηφιστεί χωριστά. Ναι, ναι, με συγχωρείτε. Υπάρχει ακόμη η τροπολογία 9 που αναφέρεται στο άρθρο 117. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 4. Για, να, για χωριστή ψηφοφορία σε τέσσερα τμήματα. Πρώτο τμήμα, ποιος είναι υπέρ. κατά αποχές εγκρίνεται με μία αποχή. Δεύτερο τμήμα, ποιος είναι υπέρ. Κατά Απορρίπτεται. Τρίτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τρίτο και τελευταίο τμήμα. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. αποχές, μία αποχή, εγκρίνεται και το τέταρτο τμήμα. Περνάμε στην τροπολογία 6 σχετικά με το άρθρο 131. Υπάρχει μία προφορική τροπολογία που προτείνει ο εισηγητής. και μπορούμε να ψηφίσουμε. Όποιο είναι υπέρ παρακαλώ να σηκώσει το χέρι του. Κατά. Αποχές. Με μία αποχή εγκρίνεται. Τροπολογία 3. Υπέρ παρακαλώ σηκώστε χέρια. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Και έτσι ολοκληρώσαμε αυτό το βαρετό έργο και μπορούμε ε, να πάμε με έτοιμο το πρόγραμμά μας εις ε, την ε, Ολομέλεια. Έκθεση Ζεύκα. Ψάχνω τον αριθμό. Λοιπόν, το σημείο 7 για την καλύτερη νομοθεσία. Κύριε Ζεύκα, θέλετε να μας σκιαγραφίσετε το περιεχόμενο της έκθεσής σας για τη βελτίωση της νομοθεσίας 15η ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 9 του πρωτοκόλλου για την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και αναλογικότητας. Δεν είναι εδώ ο κύριος Ζεύκα, αλλά νομίζω ότι παρόλα αυτά θα έπρεπε να ψηφίσουμε κύριε Πρόεδρε. δεν να προχωρήσουμε κατευθείαν στην ψηφοφορία. Allora procediamo senz'altro al voto. Προχωράμε στην ψηφοφορία. Ε, τροπολογία 5 ραονζέλ. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 4 Γιαννάκου. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 7 Χέφνερ. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Ε, τροπολογία 6 Ρονζέλ. υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 8 Ρονζέλ. ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 9 Μέσερ Σμιτ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 3, ε, τροπολογία μέσα, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται ε, 11 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 1. Χέφνερ υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Με ομοφωνία. Τροπολογία 2. Μέλτζερ. Υπέρ. Τροπολογία 2. Ανδρέας Μέλτζερ. Ωραία, είναι μόνο γλωσσικό. Οπότε εγκρίνεται διαβοής για λογικούς εύλογους λόγους. Τροπολογία 3 Hefner, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Οπότε έχουμε μόνο την τελική ψηφοφορία επ' αυτής της νομοδοτήσης όπως τροποποιήθηκε υπέρ, κατά, αποχές για να κάνουμε έναν έλεγχο πώς είναι αντίθετη. Κανείς. Άρα εγκρίνεται εκτός του κυρίου Μέσερσμιτ ε, εγκρίθηκε. Μου φαινόταν περίεργο να μην υπάρξει καμία αντίρρηση. Sarebbe un'iniziativa dei cittadini. Eh, λοιπόν, σήμερα το απόγευμα έχουμε ακόμη μόνο 5 της ημερησίας διατάξεως που αναφέρεται στην πρωτοβουλία των πολιτών ακούσαμε, μάλλον εσείς ακούσατε, γιατί εγώ τότε ήμουνα μπλοκαρισμένος από το σύννεφο της Ισλανδίας στη Ρώμη, την παρέμβαση του Επιτρόπου Σεύκοβιτς και καθορίσαμε δύο εισηγητές, τους συναδέλφους Λαμασούρ και Γκουρμάη. Και τώρα πρέπει να γίνει μία συζήτηση. Θα δώσω λοιπόν το λόγο ή στους ε, δύο μιλητές, πρώτα τον κύριο Λαμασούρ, ο οποίος μπορεί να λάβει τον λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συντονιστές και την Επιτροπή των Συνταγματικών Υποθέσεων που με ονόμασαν έναν από τους δύο συνεισηγητές παρόλη την ε, έλλειψη πείρας μου, εμπειρίας μου στην Επιτροπή σας από την αρχή αυτής της νομοθετικής θητείας. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι όπως είπατε κύριε Πρόεδρε, είχαμε μία πρώτη ανταλλαγή απόψεων κατά την ακρόαση του Επιτρόπου Σεύκοβιτς στο Στρασβούργο Ατυχώς ένας αριθμός συναδέλφων απουσίαζαν λόγω των δραστηριοτήτων του ηφαιστείου στην Ισλανδία και νομίζω ότι καλό θα ήταν σήμερα το απόγευμα να είχαμε ε, τη δυνατότητα να έχουμε μία πιο ενδελεχή συζήτηση διότι η κυρία Γκουρμάη που είχε προεδρεύσει στο Στρασβούργο τη συνεδρίαση πολύ επιτυχώς θα μπορέσει να συμβάλλει σημαντικά. Θα ήθελα λοιπόν καταρχήν να σας υπενθυμίσω το πνεύμα με το οποίο η συνταγματική συνέλευση ε, σκέφτηκε αυτή την πρωτοβουλία των πολιτών και τα, θέματα ε, ε, τα θέματα αυτά έτυχαν επεξεργασίας είτε μέσα στη συνέλευση είτε εκτός και τίθενται ορισμένα ερωτήματα επί των οποίων όλοι οι ευρωβουλευτές θα χρειαστούν την γνωμοδότηση της Συνταγματικής Επιτροπής και της, της ε, Επιτροπής Αναφορών. Πρόκειται λοιπόν για έναν τριπλό στόχο αυτών, το, αυτής της πρωτοβουλίας. Καταρχήν να υπάρχει μία έμεση διασύνδεση μεταξύ των πολιτών και των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, των Βρυξελών όπως ονομάζονται. Η ανάγκη λοιπόν αυτής της άμεσης επαφής μεταξύ των υπευθύνων για τις αποφάσεις και των αποδεκτών των αποφάσεων που είναι αισθητή σε όλα τα κράτη-μέλη, είναι πολύ αισθητή σε κοινοτικό επίπεδο διότι υπάρχουν περίπλοκες διαδικασίες παρόλη την απλοποίηση στην οποία αποσκοπεί η συνθήκη της Λισαβόνα και ε, προβληματίζουν και τα 500 εκατομμύρια πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης γι' αυτό και χρειάζεται άμεση δημοκρατία. Εμείς στην Επιτροπή είχαμε προτείνει διάφορες μεθόδους, η μόνη όμως η οποία έγινε δεκτή ομόφωνα ήταν αυτή στη συνέλευση. Δεύτερον, ο στόχος είναι να έχουν οι πολίτες την ίδια δυνατότητα πολιτικής πρωτοβουλίας που έχει και το Συμβούλιο Υπουργών και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ο καθένας μόνος του. Διατυπώσαμε λοιπόν το άρθρο αυτό με τον ίδιο τρόπο όπως το αντίστοιχο άρθρο για τις εξουσίες πολιτικής ε, πρωτοβουλίας που δίνεται από τη συνθήκη της Ρώμης στο Συμβούλιο Υπουργών και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και που τώρα επεκτείνεται στους πολίτες. Νομικά ε, η πρωτοβουλία μπορεί να έρχεται μόνο από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά η πολιτική πρωτοβουλία ε, ε, όπως αποδεικνύεται και από τις στατιστικές ε, είναι μοιρασμένη κατά εν τρίτον μεταξύ Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Κοινοβουλίου που η Επιτροπή έχει μόνο την, ε, το την νομική πρωτοβουλία ε, νομοθεσίας ε, και δεν μπορεί να υπάρξει απόφαση προτού υπάρξει ένα νομοσχέδιο που θα υποβληθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και ο τρίτος στόχος είναι να εξαλείψουμε τα τυχώματα ε, μεταξύ των πολιτικών συζητήσεων που υπάρχουν ακόμη μετά από πολλά χρόνια ευρωπαϊκής οικοδόμησης. Όλους, ε, όλα τα τείχη τα έχουμε καταλύσει εκτός από τα στεγανά των πολιτικών συζητήσεών μας. Όταν λοιπόν κατά πέντε έτη έχουμε ε, τις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βλέπουμε ότι δεν έχουμε ε, μία συζήτηση ευρωπαϊκή αλλά 27 εθνικές αμφισβητήσεις σε ένα ευρωπαϊκό σύνολο. Εάν λοιπόν υπάρξουν επαρκείς πολίτες οι οποίοι θα συμβάλλουν σε αυτή την πρωτοβουλία την ευρωπαϊκή, ελπίζουμε ότι θα υπάρξει πραγματικός ευρωπαϊκός διάλογος και τα στεγανά θα εξαφανιστούν. Ε, τίθενται όμως διάφορα θέματα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε διατυπώσει μία πράσινη βίβλο, τις οποίες ο κύριος Χέφνερ και τα δίκτυα με τα οποία συνεργάζεται ε, συνέβαλαν ε, θετικά στην επεξεργασία τους και διαπιστώσαμε ότι τίθενται πολλά πρακτικά προβλήματα. Κάθε φορά λοιπόν που έχουμε προσφυγή ή στην άμεση δημοκρατία βλέπουμε ότι υπάρχει ε, ένα πολύ εκρηκτικό θέμα σαν η τροκλικερίνη. Δηλαδή καλό είναι να απευθύνεται κανείς στο λαό εάν ελέγχεται το σύστημα αλλά είναι ε, κάκιστο εάν δεν υπάρχει ο έλεγχος αυτός διότι αντί για νητρογλυκερίνη θα έπρεπε να μιλήσω για πυρηνική ενέργεια. Δηλαδή, ε, ε, υπό τη μία, ε, υπό τη μία μέθοδο η πυρηνική ενέργεια δημιουργεί ηλεκτρισμό, υπό την άλλη έκρηξη. Λοιπόν, σε ορισμένε χώρες υπάρχει καλή χρήση, διότι ορισμένες χώρες έχουν μια δημοκρατίας όπως η πυρνική ενέργεια δημιουργεί ηλεκτρισμό ή υπό ενεργεια δημιουργει ηλεκτρισμο υπο την αλλη εκρηξη λοιπον σε ορισμενες χωρες υπαρχει καλη χρηση διοτι ορισμενες χωρες εχουν μια πολυ πλουσια εμπειρια αμεσης δημοκρατιας οπως η ελβετια και ορισμένα κράτη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως χρησιμοποιούν τα δημοψηφίσματα είτε ε, για την έγκριση νόμων ή για κατάργησή τους ή για άλλα θέματα αλλά έχουμε και πολλές περιπτώσεις σε πολλές δικτατορίες όπου η άμεση δικτατορία έχει ενισχύσει τις δικτατορίες. Λοιπόν, όλα εξαρτώνται από τον τρόπο με τον οποίο θα οργανώσουμε τη διαδικασία πρέπει να βρούμε προστατευτικά μέτρα επαρκή ώστε το δικαίωμα εκφράσεως και προτάσεως των πολιτών να λειτουργεί ικανοποιητικά σύμφωνα με το πνεύμα και το γράμμα των συνθήκων και να αποφύγουμε διαδικασίες να επιτρέψουν μία παράκαμψη της ε, ορθής διαδικασίας όσον αφορά του στόχους της συνθήκης ή κάποιας διαδικασίας που θα εμπόριζε το ε, δικαίωμα πρωτοβουλίας των, πολιτικών, των πολιτών να μπορέσει να εξασκηθεί ε, λόγω προσκομμάτων. Υπάρχουν λοιπόν διάφορα θέματα επί των οποίων θα ήθελα τη γνώμη των συναδέλφων, καταρχήν και απαριθμό εντάχει. Η συνθήκη λέει ότι χρειάζονται ένα εκατομμύρια υπογραφές, χωρίς όμως να λέει ε, πόσα κράτη-μέλη ε, θα πρέπει να έχουν προσυπογράψει την πρωτοβουλία. Λέει ένα σημαντικός αριθμός κρατών μελών. Τι θα πει σημαντικός αριθμός. Η προηγούμενη θητεία είχε ψηφίσει μία γνωμοδότηση και είχε σκεφτεί ένα τέταρτο των κρατών μελών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιστεύει το 1 τρίτο των κρατών και είναι ένα θέμα που πρέπει να εξετάσουμε. Δεύτερον, ποια είναι η ελάχιστη ηλικία για να μπορέσει κανείς να προσυπογράψει μία τέτοια αίτηση, μια τέτοια πρωτοβουλία των πολιτών, διότι η, ηλικία του εκλογικού δικαιώματος δεν είναι ίση παντού και χαμηλότερη στην Αυστρία. Δηλαδή, ε, πρόκειται να αναφερθούμε στην ε, ηλικία που χρειάζεται ε, ανακράτος για να υπογραφεί αυτό το έγγραφο ή παντού θα ισχύσει η ίδια ηλικία, οπότε θα ισχύσει το 18ο ο έτος όπου οι Αυστριακοί θα βρίσκονται σε μια ιδιαίτερη κατάσταση, 16 χρονών θα ψηφίζουν, 18 θα υπογράφουν ή θα θεωρήσουμε ότι παντού θα ισχύσει η ηλικία 16 ετών Οπότε όμως υπερβαίνουμε τη δυνατότητα πολιτικών δικαιωμάτων και εξασκήσεώς τους σε περισσότερα κράτη-μέλη. Τρίτο θέμα, το οποίο ίσως είναι το πιο δύσκολο και το πιο σημαντικό ποια στιγμή θα παρέμβει το, η εξέταση της νομικής αποδεκ, δυνατότητας αποδοχής της πρωτοβουλίας και ποιος θα προβεί σε, αυτό, σε αυτή την εξέταση. Και στο σημείο αυτό η πρόταση Κάουφμαν και Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν με ικανοποιούν. Διότι αυτός ο έλεγχος της αποδεκτικότητος της παραδοχής θα γίνει άπαξ και υπάρχει ένα ελάχιστο 10% ατόμων θα πρέπει να γίνει από την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από ένα δικαστικό οργανισμό όπως το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, από ένα ιδιωτικό ε, ιδιαίτερο θεσμό ο οποίος θα πρέπει να αποφασίσει. Πιστεύω ότι αυτό το σημείο είναι το πλέον λεπτό για να αποφασιστεί στη διαδικασία αυτή. Μετά, η συλλογή των υπογραφών η συλλογή των υπογραφών βέβαια θα πρέπει αυτοί που υποκινούν την κίνηση να φροντίσουν να μαζέψουν το ένα εκατομμύριο ε, υπογραφών. Ποιος όμως θα ελέγξει τις υπογραφές αυτές και υπό ποιες μορφής θα πρέπει να είναι ηλεκτρονικές σε χαρτί αναπτύσσεται η νέα τεχνολογία και υποθέτω ότι θα δεχθούμε τις ε, ηλεκτρονικές υπογραφές αρκεί να μπορούν να επαληθεύονται διότι στο σύντομο παρελθόν υπήρξαν αιτήσει ε, ε, ενός εκατομμυρίου υπογραφών και που ουσιαστικά βασιζόντουσαν σε 10 άτομα τα οποία είχαν χειραγωγήσει την ε, πληροφορική. Επίσης, ποιος θα πληρώσει ε, για την εργασία αυτή και ποιος θα προβαίνει στον έλεγχο, γιατί αν υπάρχει μία εθνική αρχή, μπορεί η εθνική ή περιφερειακή αρχή να είναι μαζί με, είναι με το μέρος αυτών οι οποίοι προβαίνουν στην πρωτοβουλία ή κάποιος ο οποίος είναι αντίθετός τους και θα ψηρήσει και τις λεπτομέρειες. Πιστεύω όμως ότι πολλοί συνάδελφοι ε, θεώρησαν ότι ήταν σημαντικό κατά τη συζήτηση στο Στρασβούργο ότι θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ο αριθμός των υπογραφών που θα συγκεντρώνεται σε κάθε χρόνια. Δηλαδή, αν υπάρχουν τρεις ε, υπογραφές σε μία χώρα δεν επαρκεί και το μήνυμα αυτό θα είναι το ίδιο σε όλες τις χώρες, θα διαφέρει. Ορισμένοι έχουν μαθηματικές περίπλοκες ε, σκέψεις και τους έχουμε ακούσει με μεγάλη προσοχή. Όσον αφορά τις ε, προθεσμίες, ποιες είναι οι προθεσμίες οι οποίες ε, είναι απαραίτητες για να συγκεντρωθούν αυτές οι υπογραφές με ανησυχίες αντιφατικές. Δηλαδή, ε, ένα εκατομμύριο υπογραφές χρειάζεται σε ορισμένες χώρες αρκετό χρόνο. Πρέπει όμως να σκεφτούμε και το momentum, δηλαδή το, ε, την όθηση. Ε, Ότι υπάρχει κάποια στιγμή που ξεκινά μία διαδικασία, δεν μπορεί να περιμένει κανείς τρία χρόνια για να λειτουργήσει το σύστημα αυτό. Έκτο σύστημα, πιο απλό. Ποια, το θέμα ποια θα είναι η επιπτώσεις πολιτικά και πώς θα οργανωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Διότι εφόσον η διαδικασία εξασφαλίσει ότι συγκεντρώνονται οι πολιτικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις για να αναλάβει την πρωτοβουλία Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να δούμε πώς θα προχωρήσει. Και ένα έβδομο θέμα που πρέπει να μας απασχολήσει είναι ποιες θα είναι οι λύσεις ε, ε, της οπισθοφυλακής θα μπορούσα να πω που θα μπορούσαν ε, να προταθούν ή στους υποκινητές τέτοιων πρωτοβουλειών εάν διαπιστωθεί ότι υπάρχει ενδιαφέρον πολιτικό είναι ένα ουσιαστικό θέμα το οποίο ενδιαφέρει όλους το οποίο όμως δεν συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις για να μπορέσει να εποφεληθεί της, ε, ε, ε, της σωστής διαδικασίας, δηλαδή ένα εκατομμύριο υπογραφές οπότε επιλαμβάνεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή αν είναι ένα περιφερειακό θέμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν δεν θέλουμε να έχουμε πολλούς παραπονεμένους ή όπου μόνο 10% των πρωτοβουλειών θα γίνονται αποδεκτές και το 90% θα πηγαίνει στα σκουπίδια, θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο με τον οποίο να λάβουμε υπόψη αυτές, αυτά τα διαβήματα και να δούμε ότι κάποιος τα εξετάζει. Και αυτός ο κάποιος θα είναι ποιος. Θα είναι η Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο Ευρωπαϊκός Διαμεσολαβητής, ο Εθνικός Διαμεσολαβητής, με ένα ε, ε, κατά περίπτωση θεσμικό όργανο πότε και πώς εφόσον δεν το προβλέπει η συνθήκη δεν είναι κάτι που είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε αλλά πολιτικά θα ήταν σκόπιμο να το εξετάσουμε. Όγδο θέμα τώρα. Ποιος είναι σε αυτή τη διαδικασία ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πρέπει να έχει κάποιον ρόλο. Δεν προβλέπεται από ότι συνθήκη, διότι ούτως ή άλλως το Κοινοβούλιο θα συζητήσει τα θέματα αυτά και ε, θα αποφανθεί στο τέλος. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ξεκινήσει, θα θεωρήσει ότι είτε αυτή η πρωτοβουλία των πολιτών όντως χρειάζεται ε, μία νομική συνέχεια, να διατυπωθεί δηλαδή ένα νέο κοινοτικό κείμενο ή ε, μία βελτίωση ή κατάργηση κάποιου, κάποιες νομοθεσίες ε, ή εάν ε, υπάρχει ένα πρόβλημα που δεν χρειάζεται ενέργεια θα μας το αναφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα μπορέσει το Κοινοβούλιο να το συζητήσει για να επαληθεύσει ότι έχει δίκιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά ενδέχεται να ε, γνωμοδοτήσει λέγοντας ότι ε, δεν έπραξε σωστά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αναλαμβάνοντας ορισμένες από αυτές τις πρωτοβουλίες. Δηλαδή κάποια στιγμή θα εμπλακεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και κάποια στιγμή θα συμμετάσχει στην τελική απόφαση που πρέπει να ληφθεί. Καθόλου όμως αυτή τη διαδικασία, αν δούμε ότι ορισμένα στάδια είναι πολύ σημαντικά για την επιτυχία της πρωτοβουλίας, θα χρειαστεί να λάβει, να ασχοληθεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παραδείγματο χάρη στην εξέταση του παραδεκτού της πρωτοβουλίας, ε, κατ' εμέ όχι υποχρεωτικό. Το ίδιο όμω πρέπει να αναρωτηθούμε και για τα εθνικά κοινοβούλια, όταν ε, θα ε, συγκεντρωθούν υπογραφέ, όταν θα εξεταστεί το παραδεκτό της πρωτοβουλίας μήπως κάπου θα χρειαστεί μία γνωμοδότηση εθνική του Κοινοβουλίου ή της κυβέρνηση ή του διαμεσολαβητή. Είναι ερωτήσεις που πρέπει να θέσουμε. Και τέλος το θέμα είναι του πότε θα ισχύσει το χρονοδιάγραμμα που θα καθορίσουμε για την ισχύ αυτού του νέου μηχανισμού. Ακούσαμε ότι η Ευρωπαϊκή ε, Πρωτοβουλία ενδιαφέρεται πάρα πολύ για την πρωτοβουλία των πολιτών και να θυμηθούμε ότι ο πρόεδρος Φελίπε Γκοζάλες στην αρχή της δεκαετίας του 90 είχε επιμείνει πολύ κατά τρόπον ώστε η αρχή της, ε, του ευρωπαϊκού πολίτη, ευρωπαίου πολίτου να περιληφθεί στην ε, Ευρωπαϊκή Συνταγματική Συνέλευση και θα έπρεπε ίσως να υπάρξει μία πρώτη ενδεικτική ανάγνωση και μία ψηφοφορία στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πριν από το τέλος Ιουνίου αλλά πιστεύω ότι δεν πρέπει ε, να ε, βιαστούμε πάρα πολύ. Καλύτερα το σύστημά μας να το έχουμε σκεφτεί καλά, να το έχουμε εξετάσει από όλες τις πτυχές, ακόμη και αν πάρει δύο-τρεις μήνες παραπάνω, παρά να ε, κάνουμε κάτι τσαπατσούλικο, διότι η πρώτη ανάγνωση μπορεί να γίνει αποδεκτή τον Ιούνιο από το Συμβούλιο και εμείς να έχουμε περισσότερο χρόνο, διότι αυτό το κείμενο μπορεί μπορεί να δικαιολογήσει δύο αναγνώσεις σε κάθε ένα θεσμικό όργανο προτού τελεσφορήσει. Θα πρέπει δηλαδή το σύστημα να μπορέσει να λειτουργεί στο 2011 για τις πρώτες πρωτοβουλίες πολιτών χωρίς όμως να βιαστούμε υπερβολικά. Γενικώ πιστεύω ότι η Επιτροπή ε, των Συνταγματικών Υποθέσεων ζήτησαν και την γνωμοδότηση της ε, ΟΚΕ και της Επιτροπής Περιφερειών και θα πρέπει αυτή τη στιγμή να εξετάσουμε εάν είναι κάτι το οποίο θα το συζητήσουμε στα, Ευρωπαϊ... στα Εθνικά Κοινοβούλια και πώς με μία συγκεκριμένη ε, συνάντηση των επιτροπών που είναι οι ομόλογοι μας στα Εθνικά Κοινοβούλια ή θα πρέπει να λάβουμε όλες τις προφυλάξεις για να ξέρουμε ότι θα έχουμε όλες τις αναγκαίες γνωμοδοτήσεις και οι προτάσεις τις οποίες θα κάνουμε από κοινού με την Επιτροπή Αναφορών ή στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου είναι προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις αυτής της πολύ σημαντικής και πολύ λεπτής διαδικασίας. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ για την εισήγηση. Η κυρία Γκούρμα, η αντιπρόεδρος, έχει το λόγο για τις παρατηρήσεις της. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητέ κύριε Συνεισηγητά, <clears throat> πιστεύω ότι το κοινό μας αυτό έργο μπορεί να αποδείξει ότι η συνεργασία των δύο ομάδων μας μπορεί να αποδώσει. Χαίρομαι που ο κύριος Χέφνερ θα ασχοληθεί ως ε, εισηγητής γνωμοδότησης από την Επιτροπή Αναφορών. Θα συναντηθούμε την Πέμπτη για πρώτη φορά και θα κάνουμε μια ξεκάθαρη συζήτηση για την εξέλιξη του θέματος. Ελπίζω πρώτη ανάγνωση να γίνει στη διάρκεια της Ισπανικής Προεδρίας. Συμφωνώ όμως με τον κύριο Λαμασούρο ότι αυτό που προέχει είναι δουλειά να γίνει καλά. Όπως είπε και ο Χωσέ Σαραμάγκο, οι πολίτες έχουν καθήκον να παρεμβαίνουν Δίνουμε λοιπόν την ευκαιρία αυτή στους Ευρωπαίους πολίτες με την πρωτοβουλία αυτή, που αποτελεί και σημαντική καινοτομία της ε, συνθήκης της Λισαβόνας για την ενίσχυση της άμεσης δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και βέβαια και ο συνεισηγητής μου τα εξήγησε αυτά. Ευχαριστώ όλες και όλους που μου δώσατε την ευκαιρία να συνεργαστώ για το σημαντικό αυτό θέμα. Ναι, ευχαρίστηση διεύθυνα τη συζήτηση στο Στασβούργο και βέβαια ο Σεύκοβιτς και η ομάδα του έκαναν πολύ καλή δουλειά. Είμαι βεβαία ότι με όλα αυτά στείλουμε μια γερή βάση για την περαιτέρω εργασία. Και αν είμαστε τυχεροί να έχουμε και το ψήφισμα του προηγούμενου Μαΐου και την έκθεση της Σίλβια Κάουφμαν που είναι πολύ σημαντικά ως βάση. Βέβαια, το Συμβούλιο δεν έχει συμφωνήσει. Πάντως, μία από τις διαφορές σχετικά με τον ελάχιστο ρυθμό χωρών μελών, όπως είπε και ο Ισλαμασούρ, η Κομισιόν λέει ένα τρίτο, το Κοινοβούλιο λέει ένα τέταρτο. Υπάρχει και μία μικρή διαφορά σχετικά με τον ελάχιστο ρυθμό των υπογραφών. Άλλο σημαντικό είναι το παραδεκτό της πρωτοβουλίας. Άλλη διαφορά δηλαδή. Θα πρέπει ε, να το εξετάσει αυτό η Επιτροπή μετά από συλλογή 300.000 υπογραφών. Αυτό σημαίνει βέβαια πολλή δουλειά για αυτούς που συλλέγουν τις υπογραφές που θα κάνουν την προσπάθεια αυτή και βέβαια θα θέλουν να γίνει αποδεκτή πρωτοβουλία, να γίνει παραδεκτή η πρωτοβουλία και είναι το σωστό να ψάξουμε να βρούμε τις πιο ευφυείς λύσεις για το πρόβλημα αυτό. Για τους πολίτες πρέπει να εξασφαλίσουμε ώστε η συνέχεια που θα δοθεί στην πρωτοβουλία δεν θα είναι ε, υπερβολικά μακρά και χρονοβόρα. Οι τρεις μήνες που προτείνει το ψηφισμά μας θεωρώ ότι είναι εύλογη προθεσμία. Υπάρχουν και ορισμένα θέματα τα οποία δεν έχουν διευκρινιστεί στις προτάσεις της Κομισιόν. Ας τα δούμε αυτά. Η ακρόαση των ε, οργανώσεων από την Επιτροπή. Πρέπει να δοθούν απαντήσεις εδώ γιατί υπάρχουν ορισμένα εκκρεμή θέματα την αρχή της διαδικασίας αυτής, για να πάει όμαλα, μπορούμε να στοχεύσουμε σε ορισμένα από τα σημεία αυτά της διαδικασίας. Πιστεύω ότι ο χρονικός περιορισμός δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε επιδείνωση του τελικού αποτελέσματος και πρέπει να αναζητήσουμε κοινή θέση και με τις απαραίτητες αμοιβέ παραχωρήσει ώστε το Κοινοβούλιο να μπορέσει να παίξει το ρόλο του, δηλαδή να υπερασπιστεί τι θέσει του στη διαπραγματεύση με το Συμβούλιο Υπουργών. Θα ήθελα βέβαια να ακούσω τώρα την άποψή σα, γι' αυτό βρισκόμαστε άλλωστε εδώ. Θα ήθελα να ακούσω τι υποδείξει σα για τα θέματα που ανέφερα προηγουμένω ή για άλλα σχετικά θέματα. Γι' αυτό λοιπόν θέσατε παρακαλώ υπόψη μας το τι πιστεύετε. Θεωρώ όπως άλλωστε και ο συνάδελφός μου είπε προηγουμένω, σχετικά δηλαδή με το παραδεκτό, σχετικά με την συλλογή των υπογραφών, ότι πρέπει να γίνει συζήτηση. α είμαστε όμω, α μείνουμε όμως στα όρια της λογικής συζήτησης και σε συνεργασία βέβαια με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με τον Επίτροπο Σεύκοβιτ, που έχει δείξει πνεύμα συνεργασίας μαζί μας. Θα ακούσω λοιπόν με ε, μεγάλη χαρά της απόψεις. Ευχαριστώ λοιπόν και τον συνεταίρο μου, τον εισαγωγικών, τον κύριο Ραμασούρ και εσάς βεβαίως κύριε Πρόεδρε. Για την Επιτροπή Αναφορών, ο κύριος Χέφνερ έχει το λόγο. Του δίνω λοιπόν το λόγο πρώτου και καλύτερο. Σα Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Πρώτα, επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω ε, τους κύριους Λαμασούρ και Γκούρμαϊ για την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα εισαγωγή στο θέμα που δείχνει ότι υπάρχει κοινή αντιμετώπιση και σε ό,τι αφορά τις δυνατότητες που μας ανοίγονται αλλά και σε ό,τι αφορά τα καθήκοντα, τις υποχρεώσεις που προκύπτουν για μας, στα πλαίσια δηλαδή της συμμετοχής του Κοινοβουλίου στην νομοθετική διαδικασία. Όχι μόνο στο Στρασβούργο συναντηθήκαμε με τον ε, Επίτροπο Σεύκοβιτς για να συζητήσουμε το θέμα αυτό. Προηγουμένως είχε κάνει η Επιτροπή διαδικασία διαβουλεύσεως και στις 22 Φεβρουαρίου είχε διοργανώσει μεγάλη ακρόαση με συμμετέχοντες της κοινωνίας των πολιτών, όπου εγώ είχα την τιμή να εκπροσωπήσω την παρούσα επιτροπή. Το λέω αυτό διότι υπάρχει μια σύνοψη της Ακρόασης αυτής από πλευρά κομισιών και μια συνολική επισκόπηση των προτάσεων που έγιναν. Όσοι επιθυμούν εδώ να εγκύψουν στο θέμα, ας την εξετάσουν. Υπάρχουν, περιλαμβάνονται σε αυτή τη σύνοψη, πολλές ενδιαφέρουσες σκέψεις. Επίσης, η ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών διεξήγαγε προ δύο εβδομάδων περίπου μια σχετική ε, συνεδρίαση και η ομάδα των Πρασίνων διοργανώνει παρόμοια για την επόμενη εβδομάδα στις 12 Μαΐου. Θα γίνει το απόγευμα και είστε όλοι βεβαίως εγκαρδίως προσκεκλημένοι. Νομίζω ότι θα πρέπει και ως Επιτροπή να κάνουμε το ίδιο, δηλαδή να προσκαλέσουμε και εμπειρογνώμονες αλλά και τους λεγόμενους stakeholders, δηλαδή τους ενδιαφερομένους και συμφωνώ επομένω με την διατύπωση του Αλάν Γαμασούρ. Εγώ θα το έλεγα με τα δικά μου λόγια ως εξή να προχωρήσουμε με ταχύτητα αλλά όχι με βιασύνη. Πιέζει ο χρόνο, αλλά χρειαζόμαστε μια στέρεα νομοθεσία. Γι' αυτό ας προχωρήσουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα. Δεν θα μπω σε πολλές λεπτομέρειες. Ίσως μερικά βασικά. Στην πυρήνα, στον πυρήνα του μάλλον το θέμα είναι να επιτραπεί στους πολίτες να ζήσουν πραγματικά αυτή την Ευρώπη, όχι μόνο δια της ψήφου των, όχι μόνο με τη συμμετοχή τους εκλογές, αλλά ε, ότι ε, τους ανοίγεται η πόρτα και να συμμετάσχουν άμεσα. Δηλαδή υπάρχει εδώ στις Βρυξέλλες μια πόρτα ανοιχτή για τους πολίτες για να μπορέσουν να υποβάλουν τα αιτήματά τους για να μπορέσουν να υποβάλουν προτάσεις. Έτσι εγώ δεν θα τόνιζα πρώτα-πρώτα τους κινδύνους. Συμφωνώ ότι υπάρχουν βέβαια κίνδυνοι, αλλά η ευφία του νομοθέτη πρέπει να είναι να αποφύγει τις κοπέλους και θα το έλεγα ίσως πιο οξυμένα ότι είναι λιγότερη κινδυνική από ότι είναι η κίνδυνη στην, κοινωνία, στην πρωτοβουλία των πολιτών, δηλαδή από την κίνδυνη των χρηματαγορών. Μπορούμε λοιπόν να βάλουμε ρήτρε που να αποτρέπουν οποιαδήποτε κατάχρηση. Εν τέλει, ο κίνδυνο θα είναι μεγαλύτερο αν δεν υπάρξει η πρωτοβουλία των πολιτών. Γιατί ο κίνδυνο που διαβλέπω εγώ είναι να απολέσουν ενδιαφέρον οι πολίτε, να αποστρέψουν το πρόσωπό του από την Ευρωπαϊκή Ένωση και επομένω εν τέλει να απολέσει αξιοπιστία η Ένωση. Εδώ τους ανοίγεται ένας δρόμος ο οποίος τους επιτρέπει να θέσουν θέματα και με τη διαδικασία αυτή μπορούν να απτυχθούν ιδέες και να προταθούν ή και να απορριφθούν. Γιατί η πρωτοβουλία των πολιτών μπορεί ε, να έχει και το νόημα ότι εμείς οι πολίτες δεν θέλουμε να προχωρήσει η τάδε ιδέα. Πάντως θεωρώ ότι πρόκειται για μεγάλη πρόοδο, μεγάλο βήμα πρόοδου για την Ευρωπαϊκή Ένωση και χαίρομαι που μπορούμε να προχωρήσουμε να την καταστήσουμε ισχύον δίκαιο. Για τα επιμέρους θέματα που τίθενται, θα ήθελα να τονίσω ιδιαίτερα δύο. Αφενός, περί τα αντικείμενα. Κάπου μένει κρυμμένο νομίζω ότι ακόμα δεν έχει γίνει πλήρης η διατύπωση του σχετικού κειμένου. Δηλαδή, άλλωστε το είπε και ο κύριος Λαμασούρ προηγουμένως και υπενθυμίζω ότι όσοι είχαν συμμετάσχει τότε στην συνέλευση όπως Λαμασούρ, Φόκεν, Χούμπερ και άλλοι είχαν υποστηρίξει την ιδέα αυτή, έχοντας πάντοτε υπόψη ένα παραλληλισμό με τις δυνατότητες που δίνει η συνθήκη της Λισαβόνας και στο Συμβούλιο Υπουργών και στο Κοινοβούλιο να υποβάλουν τέτοιου είδους προτάσεις. Αυτό όμως βέβαια ανοίγει και το θέμα πώς και από ποιον μπορεί να κρυθεί τι είναι παραδεκτό και τι όχι. Εδώ θεωρώ ότι πρέπει να βασανίσουμε τα κύτταρα του εγκεφάλου μας, γιατί νομίζω ότι δεν έχει δοθεί ακόμα τελική λύση σε αυτό. Ε, το όριο των 300.000 υπογραφών μου φαίνεται ότι καθυστερεί πάρα πολύ. Εχετε δηλαδή σε πολύ καθυστερημένη φάση. Τι είστε λοιπόν το θέμα ποιος κρίνει, με ποια διαδικασία υπάρχει δυνατότητα προσφυγής σε περίπτωση αρνητικής απόφασης. Αυτά πρέπει να απαντηθούν μέσα στα πλαίσια της έκθεσης. Τα μεγάλα θέματα τα έθιξε ο Λάλα Μασούρ στην πρώτη του τοποθέτηση. Κάποια θέματα μένουν και για το τέλος της διαδικασίας. Και μένα με απασχολεί ποιε θα είναι οι ένομε συνέπειες μια τέτοια πρωτοβουλία των πολιτών. Αυτό δεν μπορεί να μείνει ανοιχτό. Όταν λέω ένομε συνέπειε δεν εννοώ ότι η πρωτοβουλία των πολιτών έχει και την απέτηση να υλοποιηθεί, γιατί αυτό το αφήνει ανοιχτό η συνθήκη της Λισαβόνας είναι κυρίαρχη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αποφασίσει εάν θα δεχθεί την ε, πρόταση αυτή, την πρωτοβουλία αυτή, εάν θα ξεκινήσει μια νομοθετική διαδικασία ή όχι. Αλλά δεν μπορεί και δεν επιτρέπεται να μείνει ανοιχτό το πώς θα αντιδράσουν διαδικαστικά τα όργανα και ιδίως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρέπει να υπάρχει μια τακτοποιημένη διαδικασία ώστε να μην έχουν την εντύπωση αν θέλει οι πολίτες ότι ξεσηκώνονται κατά εκατοντάδε χιλιάδε, παλεύουν ένα χρόνο ολόκληρο, μαζεύουν υπογραφέ, τι στέλνουν στι Βρυξέλλε και εν τέλει ούτε, ούτε, ούτε μια σοβαρή απάντηση δεν λαμβάνουν και δεν κινείται απολύτω τίποτε. Αυτά πρέπει να μα απασχολήσουν. Πάντω, έχει υποβληθεί μια καλή πρόταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία βέβαια χρήζει βελτιώσεων, αλλά αποτελεί μια σοβαρή βάση για τη συνεργασία και νομίζω μάλιστα ότι και στην διάρκεια τη παρούσα εβδομάδα θα περάσει, θα διαβαστεί και στο Κοινοβούλιο, όχι μόνο στην Επιτροπή Συνταγματικών, που έχει κάνει ήδη το καθήκον της με τον διορισμό εισηγητών, αν και υπάρχουν και άλλοι εισηγητές που δεν έχουν διοριστεί ακόμα. Πάντως μπορούμε να αρχίσουμε τη δουλειά που νομίζω ότι ε, θα είναι ιδιαίτερα ικανοποιητική από κάθε άποψη. κύριος Μέσσερ Σμιτ. λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και ευχαριστώ και τους εισηγητές για την πολύ καλή παρουσίασή τους. Θέλω να επανέλθω στα κριτήρια, τα τυπικά και ουσιαστικά κριτήρια που αναφέρονται, αριθμό υπογραφών, χώρα προέλευσης κλπ. Αυτά είναι τα τυπικά κατά την, άποψή μου κριτήρια. Θα έπρεπε στο σημείο αυτό να έχουμε σαφείς απαιτήσει. Πιο επικίνδυνο είναι να ξεκινήσουμε να ελέγχουμε τα ζητήματα που μπορούν να εξεταστούν. Εμείς ως κοινοβούλιο είναι σαφές ότι θα έχουμε μία θέση για τις προτάσεις που θα υποβληθούν. Οι θέσεις αυτές θα πρέπει να αντικατοπτρίζονται στη διαδικασία καθοδών. Αλλά να ξεκινούμε με ε, την αφετηρία ότι μια πρωτοβουλία δεν μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλες αλλαγές και να λέμε ότι αυτό το θέμα δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί εξ αρχής. Ε, νομίζω ότι δεν είναι καλή ιδέα. Δηλαδή δεν ε, δεν στέκει. Και με ανησύχησε το ότι άκουσα τον Σεύκοβιτς να λέει ότι οι προτάσει που, πρέπει να γίνουν, που μπορούν να γίνονται εκτέ θα πρέπει να εντάσσονται σε ένα πλαίσιο. Εγώ πιστεύω ότι ε, πολλέ προτάσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσαν να πάρουν, να μαζέψουν ένα εκατομμύριο υπογραφέ και να τηρούν του όρου. Προφανώ μετά θα χρειαστεί μια πλειοψηφία στο Συμβούλιο του Υπουργών, στο Κοινοβούλιο κλπ. σω να μην υπάρξει πλειοψηφία για την πρόταση αυτή. Το ότι δεν υπάρξει πλειοψηφία ωστόσο δεν νομίζω ότι είναι σωστό να πούμε ότι επειδή δεν θα έχει πλειοψηφία δεν θα την προχωρήσουμε. Πρέπει να δώσουμε όσο μεγαλύτερη ελευθερία γίνεται στην οριοθέτηση των θεμάτων που μπορούν να πληρούν τα κριτήρια και μπορούν να προχωρήσουν. Αν δείτε τι γίνεται στην Ευρώπη, θα δείτε ότι μπορεί να βρούμε ένα μοντέλο που μπορεί να λειτουργήσει ως πηγή έμπνευση. Δεν νομίζω όμως ότι πρέπει να αναζητήσουμε κάτι τέτοιο σε μια χώρα που θα έχει παρόμοια δομή. Ε, η Ελβετία, για παράδειγμα, έχει συγκεκριμένους κανόνες. Έναν αριθμό πολιτών που μπορούν να ζητήσουν την προκήρυξη ενός δημοψηφίσματος. Εγώ δεν θέλω την ελβετική νομοθεσία, αλλά θα μπορούσαμε να δούμε τι λειτουργεί στην Ελβετία. Ποιε είναι οι τυπικέ προποθέσει και οι υλικέ προποθέσει για την διοργάνωση ενό δημοψηφίσματο και πιστεύω ότι αυτό θα μπορούσε να λειτουργήσει σαν πηγή έμπνευση. Θα μπορούσαμε να δούμε πώς λειτουργεί στην πραγματικότητα κάτι τέτοιο. Αυτό είναι το ουσιαστικό πιστεύω. Στα 27 κράτη-μέλη πιστεύω ότι υπάρχει προσδοκία από την μετατροπή της πρωτοβουλίας αυτής σε, ε, μια πραγματική, σε ένα πραγματικό μοίρασμα των αρμοδιοτήτων με μεταξύ θεσμικών οργάνων και πολιτών. Ας ψάξουμε λοιπόν στην Ήπειρο να βρούμε ποια μοντέλα έχουν μια τέτοια πρόθεση, που μπορεί να μην είναι ακριβώς ίδια. Να προσθέσω, αν μου επιτρέπετε, και κάποιες σκέψεις για τα κριτήρια που αναφέρατε. Είναι σημαντικό να υπάρχει και ένα κριτήριο αποδέκτη των προτάσεων. Αν θυμηθούμε στο παρελθόν, στην προεκλογική εκστρατεία υπήρχαν μια σειρά κλισέ, ανάπτυξη, σταθερότητα, προόδος, ωραία λόγια. Είναι λοιπόν σημαντικά να διευκρινίζουμε, να λέμε ότι η, μεταξύ των τυπικών προϋποθέσεων να υπάρχει πολύ συγκεκριμένη διατύπωση για το πώς θα επιτευχθούν οι στόχοι. Να μην έχουμε δηλαδή ένα γενικό πλαίσιο, αλλά πολύ συγκεκριμένες προτάσεις. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό να πρόκειται για δημοκρατική πρωτοβουλία και κατά συνέπεια να τηρούνται τα τυπικά κριτήρια. Να μην μιλάμε για αξίε μόνο, να μην περιοριζόμαστε μόνο στι ε, ευρωπαϊκέ αξίε, όπω είπε ο κ. Σεύκοβιτ. Πρέπει κάθε πρωτοβουλία να αντιμετωπίζουμε και να εξετάζουμε κάθε πρωτοβουλία που θα παίρνει ένα εκατομμύριο πολιτών. Κύριος Τασκόφσκι. Καταρχάς να ευχαριστήσω του τους συναδέλφους για την παρουσίασή τους. θα μιλήσω για το πιο ευαίσθητο ζήτημα κατά την απόψή μου, το θέμα του παραδεκτού. Και θέλω να πω κάτι. Είναι προφανές ότι το ζήτημα αυτό πρέπει καταρχάς να το, να το κρίνει η Κομισιόν, αν θέλουμε να διαφυλάξουμε το μονοπόλιο της πρωτοβουλίας που, ισχύει, που ισχύει στην ε, κοινοτική μέθοδο. Αυτό ε, μετά όμως τι γίνεται. Υπάρχει δυνατότητα προσφυγή στο ΔΕΚ αν θεωρούν οι συντάκτε τη πρωτοβουλία αυτή ότι πρέπει να προσφύγουν στο ΔΕΚ, τι γίνεται. Διότι μπαίνουμε σε ένα ναρκοπέδιο. Μπαίνουμε στο ζήτημα των competence competence, της αρμοδιότητας των αρμοδιοτήτων, της ε, κατανομής αρμοδιοτήτων μεταξύ εθνικών και Ευρωπαϊκού ε, Δικαστηρίου. Ο κ. Ντάφ λέει ότι δεν είναι μεγάλο το πρόβλημα, διότι το ΔΕΚ δεν θα λύσει το ζήτημα αυτό όπως έκανε με το θέμα της επικουρικότητας. Ίσως όμως και όχι. Αυτό είναι το ζήτημα κλειδί στη συζήτηση που έχουμε. Ευχαριστώ. Grazie, onorevole Guerrero. Ο κύριος Γκερέρο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κάποιες παρατηρήσεις θέλω να κάνω και κάποιες σκέψεις για να βοηθήσω τους συγγητές να ε, αντιμετωπίσουν το ζήτημα αυτό. Όπως είπε ο κύριος Λαμασούρ, πρόκειται για μια πρωτοβουλία που θέλει να σπάσει το γυάλινο τείχο που χωρίζει τους πολίτες από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Είναι λοιπόν μια πρωτοβουλία που τελειοποιεί τη δημοκρατία και την εμπλουτίζει κατά συνέπεια. Ωστόσο, πιστεύω ότι πρέπει καταρχάς να διαμορφώσουμε ένα πλαίσιο παιδαγωγικό ευνοϊκό προς την αντιπροσωπευτική δημοκρατία. Η πρωτοβουλία δεν είναι εναλλακτική λύση, αλλά συμπλήρωμα της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας. Πλουτίζει την αντιπροσωπευτική δημοκρατία. Όσο είχαμε κοινοβούλια, είχαμε δημοκρατία. Αντίθετα, δεν είχαμε πάντα δημοκρατία όταν είχαμε άμεση δημοκρατία. Πρέπει λοιπόν να έχουμε επίγνωση του ότι η βάση του πολιτικού μας συστήματος εδράζεται στην αντιπροσώπευση. Καρπός της αντιπροσώπευσης είναι βεβαίως η βούληση των πολιτών, οι οποίοι είναι αυτοί που εκλέγουν ένα κοινοβούλιο και μέσω αυτού τα άλλα όργανα. Δεν χρειάζεται λοιπόν να προασπίζουμε την σημασία της πρωτοβουλίας για την αντιπροσώπευση της ε, για, την, ε, για τον εμπλουτισμό της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας, να υπογραμμίσω ότι δεν πρόκειται για εναλλακτική λύση. Δεύτερη παρατήρηση. Τα δικαιώματα διακηρύσσονται. Εμεί, το Σύνταγμα ή στη Συνθήκη τη Λισαβόνα διακηρύξαμε το δικαίωμα των πολιτών να ασκήσουν την, από την προσωπευτική δημοκρατία. Όταν όμως ρυθμίζουμε τα δικαιώματα, τα περιορίζουμε. Πάντα θεσπίζουμε τους όρους μέσω των οποίων ασκούνται τα δικαιώματα αυτά. Τούτο γίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και οπουδήποτε αλλού σε εθνικό πλαίσιο. Ο όρος ή η προϋπόθεση είναι ότι οι περιορισμοί στα δικαιώματα δεν μπορούν να αλλοιώσουν την ουσία τους. Δεν μπορούν να οδηγήσουν το να παρεμποδίσουμε την πραγματική άσκηση του δικαιωμάτων αυτών μέσω της ε, ρύθμισής τους. Άρα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί με, τη, με τους περιορισμούς. Πρέπει ωστόσο να έχουμε επίγνωση ότι κανένα δικαίωμα δεν ασκείται εν κενό, χωρίς, νόμοθεση, χωρίς ρύθμιση και περιορισμό. Πιστεύω ότι το βασικό θέμα, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, είναι το θέμα του παραδεκτού το, για το θέμα αυτό πρέπει να είναι σαφές εξ αρχής ποιοι είναι οι περιορισμοί. Κατά άποψή μου πρέπει να είναι λίγοι, σαφείς και γνωστοί από όσους προσπαθούν την ΑΒ στιγμή να ασκήσουν το δικαίωμα αυτό σε κάποια χώρα της Ένωσης ή σε όλες τις χώρες της Ένωσης. Πιστεύω ότι πρέπει να σκεφτούμε κάποιους πιθανούς ε, περιορισμούς και λέω να σκεφτούμε γιατί δεν θέλω να δηλώσω ότι είμαι υπέρ του να θέσουμε εξ αρχής ε, περιορισμούς. Εγώ νομίζω ότι αυτό πρέπει να αφορά το περιεχόμενο των θεμάτων που θα πρέπει να αφορά η πρωτοβουλία αυτή. Να σκεφτούμε, περιφερειπή, αν είμαστε έτοιμοι να δεχθούμε σύγκρουση σαφείς περιπτώσεις σύγκρουσης ε, νομιμότητας αποφάσεων κοινοβουλίου και άμεσης νομοθετικής πρωτοβουλίας. Άμεσης. Γιατί άμεσης μπορεί να υπάρχει μια νομοθετική πρωτοβουλία πολιτών με το πέρασμα του χρόνου. Ο πρόεδρος ωστόσο έρχεται από μια χώρα δεν θα πω τίποτα για τη χώρα αυτή, γιατί εσείς πρόεδρε έχετε δεκαετίες εμπειρία στον τομέα αυτό όπου πολλές φορές το δημοψήφισμα που στην Ισπανία λέγεται, ορίζεται ως καταργητικό δημοψήφισμα, δηλαδή δημοψήφισμα που αφορά μία άμεση κοινοβουλευτική απόφαση, αποτελεί μόνιμη περίπτωση σύγκρουσης νομιμότητας και άρα ε, πολιτικής αποσταθεροποίησης. Κάτι που ενέκριναν τα θεσμικά όργανα της Ένωσης το πρώτο εξάμεινο, για παράδειγμα, του 2011, θα έπρεπε να εξετάσουμε. Είναι λογικό να έχουμε μία νομοθετική πρωτοβουλία αντίθετη με αυτό το κείμενο δύο, δύο μήνες μετά. Μήπως πρέπει να βάλουμε κάποιο χρονικό διάστημα. Μήπως πρέπει να εξετάσουμε κατά πόσο θέλουμε να υπάρχει μια σύγκρουση νομιμοτήτων της θεσμική ή αντιπροσωπευτική με την λαϊκή. Επίσης θα έπρεπε να, να εξετάσουμε, μη τυχόν θα έπρεπε να, ε, να εξετάσουμε ενδεχόμενε ε, ενδεχόμενους τους, στα λεγόμενα ηθικά διλήμματα. Να σας δώσω μια κρέα περίπτωση μία πρωτοβουλία για την θανατική ποινή. Υπέρ της θανατική ποινή. Εγώ έχω σοβαρέ επιφυλάξει για το αν θα έπρεπε να θέσουμε κάποιου περιορισμού σε τέτοια ζητήματα. cuestiones, por ejemplo, impositivas. de los impuestos. Φορολογικά ζητήματα. Εάν υπήρχε πρωτοβουλία πολιτών, προφανώς φόρος δεν θα υπήρχε πουθενά. Το ξέρουμε. Δεν λέω να μην έχουμε να, έχουμε, να απαγορεύουμε την νομοθετική πρωτοβουλία σε φορολογικά θέματα, αλλά το σκεφτούμε. Και υπάρχει και άλλο ένα θέμα που αφορά τη χρηματοδότηση. Δύσκολο ζήτημα. Όπως γνωρίζετε, Η χώρα που έχει τη μεγαλύτερη άμεση δημοκρατία δεν είναι όπως νομίζετε η Ελβετία, αλλά οι Ηνωμένε Πολιτείε. Όπου πάμπολες πολιτείε έχουν στον εκλογικό τους νόμο δεκάδες κάθε φορά, σε κάθε εκλογή έχουν δεκάδες προτάσεις ε, δημοψηφίσματος. υπάρχει ε, σημαντική βιβλιογραφία πολιτιολόγων που δείχνουν ότι στα δημοψηφίσματα αυτά, όσα περισσότερα λεφτά βάζει, τόσο ευκολότερα γίνονται δεκτά. Υπάρχει λοιπόν ο κίνδυνος έμεσα να χρησιμοποιείται η νομοθετική πρωτοβουλία για συντεχνιακά συμφέροντα, για λόμπι κλπ. Ας δούμε λοιπόν κάτι για την χρηματοδότηση. Συμφωνώ με διάφορους ομιλητές ότι η πρωτοβουλία πρέπει να έχει κάποια συνέχεια αν δεν οδηγεί σε κάτι συγκεκριμένο. Δεν είναι εύκολο να λέμε ελάτε να υπογράψετε και μετά το αφήνουμε στην άκρη. Και κάποια σχόλια για το χρονικό στοιχείο. Όπως είπε ο κ. Λαμασούρ, ότι πρέπει να σπάσουμε αυτό το γυάλινο το γυάλινο ταβάνι όσο περισσότερο χτυπάμε αυτό το γυάλινο τείχο τόσο πιο αξιόπιστοι θα είμαστε. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα σπάσει με το πρώτο, αλλά πρέπει να προχωρήσουμε παρκώς για να δώσουμε ένα μήνυμα, ένα σαφές μήνυμα, ότι αυτός ο, ξύλινο, ο γυάλινος συγγνώμη, τείχος θα σπάσει. Δεν είναι ασήμαντο το ότι αυτή τη στιγμή μπορούμε να λάβουμε την υποστήριξη της Ισπανικής Προεδρίας για να προχωρήσουμε όσο περισσότερο γίνεται. Εγώ συμφωνώ ότι είναι καλύτερο να υπάρχει μια σωστή νομοθέτηση της πρωτοβουλίας παρά μια κακή άμεση εφαρμογή. Το πολιτικό μήνυμα ωστόσο που μπορούμε να περάσουμε είναι ότι πάμε με το ίδιο βήμα προς την ίδια κατεύθυνση με την προσωρινή προεδρία του Συμβουλίου είναι ένα μήνυμα καλό που πρέπει να το εκμεταλλευτούμε. Κύριε Πρόεδρε, πρόκειται για πολύ σημαντική πρόταση που ενδέχεται να επηρεάσει και του, να καθορίσει μάλλον και του τι είδους δημοκρατία θα, θα είμαστε. Δεν είναι μόνο το χαρακτηριστικό της άμεσης δημοκρατίας. μεταφέρει τις πολιτικές που ασκούμε εδώ και στο άμεσο εθνικό πλαίσιο. Τα εθνικά πολιτικά κόμματα, δηλαδή θα εντυπωσιαστούν ασφαλώς από το πείραμα μας αυτό. Θα επηρεάσει δηλαδή τις εσωτερικές πολιτικές στις χώρες μέλη. Με έναν τρόπο που δεν θα μπορούν να ελέγξουν. Και δεν θα τους αρέσει, γιατί δεν τους αρέσει να μην έχουν τον έλεγχο των πολιτικών τους. Είναι λοιπόν απαραίτητο να φανούμε πάρα πολύ σόφρονες. Και ας μην βιαστούμε να ολοκληρώσουμε την συζήτηση αυτή πριν από το τέλος της Ισπανικής Προεδρίας. Γιατί δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο χωρίς βιασύνη. Θεωρώ την πρόταση της Κομισιόν στο σύνολό της καλή και πάντως βελτίωση ε, απέναντι στην έκθεση Kaufman. Υπάρχουν ωστόσο πλείονα θέματα που δεν έχουν τεθεί στο σχέδιο αυτό. Ο Αλάν ήδη ανέφερε ορισμένα και ας με επιτρέψει να προσθέσω μερικά ακόμη. Είναι σημαντικό να μην απογοητεύσουμε το κοινό Το θέμα του παραδεκτού, όπως αναγνωρίσαμε όλοι, βρίσκεται βέβαια στον πυρήνα του προβλήματος. Θα πρέπει να πούμε ρητά στο σχέδιο ότι η πρωτοβουλία των πολιτών θα πρέπει να εμπίπτει πλαίσια στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τη Ένωσης. Βέβαια δεν λέγεται αυτό ρητά, πρέπει να, να δεχτεί ρητά και υπάρχουν βέβαια και τριών ειδών αρμοδιότητες η αποκλειστική, η κοινή και η συμπληρωματική και αυτή κάπως ασαφής περιγραφή και ο ορισμός των συμπροβατικών αρμοδιοτήτων. Είναι γνωστό ότι υπάρχει. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να ε, διατυπώσουμε σαφώς ποια αποκλείονται και ποια όχι. Βέβαια, η αδίποτε πρωτοβουλία θα πρέπει να σέβεται τον χάρτη. Για παράδειγμα, μια πρωτοβουλία που θα προβαίνει σε έκκληση να επαναφερθεί η θανατική ποινή, τουλάχιστον κατά τη δική μου ερμηνεία, θα είναι αντίθετη στον χάρτη. Ίσως λοιπόν αυτό μπορεί να μας βοηθήσει στο να εξετάσουμε τι θα πρέπει να αποκλειστεί. Επίσης θα πρέπει να πούμε ότι θα πρέπει να είναι εντός των πλαισίων των εξουσιών των θεσμικών οργάνων, που έχουν βέβαια αυξηθεί και της Επιτροπής και του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου. Ωστόσο δεν είναι αυτονόητο ότι οι εξουσίες των οργάνων μπορούν να οριστούν με ακρίβεια. Σε ένα κείμενο του είδους αυτού. Εάν για παράδειγμα μια πρωτοβουλία πολιτών προτείνει αλλαγή της συνθήκης. Τι θα κάνουμε. Είναι λίγαν πιθανό κάποια πρωτοβουλία πολιτών να προτείνει τροποποίηση της συνθήκης. που δεν είναι καθαρά νομοθετική απόφαση των θεσμικών οργάνων, αλλά δεν είναι και πάρα πολύ μακριά. Για παράδειγμα, να ψηφιστεί μια πράξη η οποία θα ξεκινήσει την διοργάνωση μιας διακυβερνητικής διασκέψεως. Είναι ε, μια απόφαση με μεγάλη βαρύτητα, αλλά ε, θα είμαστε υπερβολικά τυπολάτρες και θα πούμε «Α, όχι, πολίτες, δεν μπορείτε να ζητήσετε κάτι τέτοιο, διότι είναι εκτός του περιεχομένου των ρήτρων. Δεν είμαι βέβαιος ότι μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Υπάρχουν και ορισμένες περιπτώσεις όπου όπου και το Κοινοβούλιο μπορεί οι ορισμένε προϋποθέσεις να αναλάβει πρωτοβουλίες εκλογική διαδικασία, για παράδειγμα. Τροποποίηση του καθεστώτος των πολιτικών κομμάτων. Τέτοια πράγματα υπάγονται σε δικαίωμα πρωτοβουλία του Κοινοβουλίου. Εάν τώρα η πρωτοβουλία πολιτών υπησέλθει σε τέτοια θέματα, απευθυνόμενοι ωστόσο στην Κομισιόν, τι θα πει τότε η Κομισιόν. Όχι, δεν μπορούμε να το αγγίξουμε γιατί δεν είναι δική μας υπόθεση. Ή μπορούμε να περιλάβουμε μια διαδικασία στο σχέδιο αυτό που θα επιβάλλει στην Κομισιόν να διαβιβάζει τέτοιου είδου πρωτοβουλία σε εμά, στο Κοινοβούλιο. Δηλαδή. Τέταρτο, νομίζω ότι η διαδικασία για τη λήψη απόφασης περί του παραδεκτού και επειδή θα είναι ιδιαίτερα αμφιλεγόμενη, θα πρέπει να διαθέτει και διαδικασία προσφυγής κατά της πρώτες αποφάσεως. Θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα δηλαδή οι άνθρωποι να παραπονεθούν απέναντι σε κάτι που δεν θα είναι ούτε το δικαστήριο ούτε ο συνήγορος του πολίτη. Ο συνήγορος του πολίτη ενδιαφέρεται πάρα πολύ για τη διαδικασία αυτή και θα προτείνω να τον προσκαλέσουμε να έλθει σε μία από τις επόμενες συζητήσεις στην Επιτροπή Συνταγματικών Θεμάτων να μιλήσουμε μαζί του γιατί έχει και συμμετοχή σε θέματα συμμετοχικής, συμμετοχικής δημοκρατίας αλλά έχει και προτάσεις που, μπορεί, που μπορούν να μας βοηθήσουν να μεταθέσουμε τέτοιες πρωτοβουλίες εφόσον προκύψουν. Τέλος, ε, στην πρόταση που κάνω για την τροποποίηση της εκλογικής διαδικασίας περιλαμβάνω δύο προτάσεις που μπορούν να μας βοηθήσουν στο να βελτιώσουμε τον κανονισμό της πρωτοβουλίας των πολιτών. Πρώτα, προτείνω την καθίδρυση μιας εκλογικής αρχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα επαληθεύει τις διαδικασίες για την εκλογή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορούν να τις ανατεθούν και εξουσίες επαληθεύσεως ενδεχομένως μιας πρωτοβουλίας πολιτών θα είναι δηλαδή ένα ιδιαίτερο όργανο το οποίο δεν υπάρχει ακόμη και θα είναι εγκατεστημένο εκτός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεύτερο, προτείνω μια ξεκάθαρη διατύπωση ε, μια αρχή φθήνουσας αναλογικότητας που μπορεί να μας βοηθήσει να ρυθμίσουμε το θέμα που έθεσε ο Ράνα Μασούρ σχετικά με τον απαραίτητο αριθμό υπογραφών για κάθε χώρα. Θα επανέλθουμε σε αυτά, ελπίζω σύντομα. Αλλά πάντως, όπως ε, είπα και προηγουμένως, προτείνω εν τέλει να προσκαλέσουμε τον Ombudsman να έρθει να συνομιλήσει μαζί μας. Ευχαριστώ, Σούλτς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ζήτησα ιδίω το λόγο διότι κατά τη συζήτηση διαπίστωσα ότι δεν ε, πρέπει να ε, καταρρύψουμε το όλο σύνολο. Δηλαδή θέλω να ευχαριστήσω και τον κύριο Χέφνερ και τον κύριο Λαμασούρ διότι περιέγραψαν το πρόβλημα επακριβώς το οποίο τίθεται ε, με την επεξεργασία της προτάσεως Ευρωπαϊκής Επιτροπής και είναι κάτι που πρέπει να αντιμετωπίσουμε πολύ σοβαρά γιατί η διατύπωση και αποδοχή αυτού, του, αυτής της δυνατότητας της συνθήκης της ε, Λισαβόνας θα επηρεάσει τους λαούς των 27 χωρών δηλαδή θα τους δώσει τη δυνατότητα να επηρεάσουν άμεσα την πολιτική ε, πολιτική ε, που επηρεάζει τους πολίτες. Λοιπόν, ε, θα πρέπει να προσπαθήσουμε να επιτύχουμε ε, να προχωρήσουμε γρήγορα και να καταστεί σαφές ότι η διαδικασία αυτή θα ξεκινήσει το 2010 με όλα τα περίπλοκα ερωτήματα τα οποία συνεπάγεται, δηλαδή ε, ποιος αριθμός υπογραφών θα ε, απαιτείται για μια τέτοια πρωτοβουλία των ε, πολιτών για να γίνει νομικά δεσμευτική. Δηλαδή, ποιες θα είναι οι παράμετροι αυτών των παραμέτρων των πολιτών με ε, πόσο θα γίνει ε, πολιτικά δεσμευτική ε, για τον εμπλεκόμενο, το εμπλεκόμενο θεσμικό όργανο. Υπάρχει το πρόβλημα της χρηματοδότησης, διότι αυτό είναι σαφές και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο και εμείς θα πρέπει ε, να αντιληφθούμε ότι θα χρειαστεί να διαθέσουμε ε, ένα ποσό για αυτές τις πρωτοβουλίες και ε, σε τι θέματα θα πρέπει να αφιερωθούν οι πόροι αυτοί, ενδεχομένως παραδείγματος χάρη και στο θέμα αλλαγής των συνθήκων για την εποπτεία των τραπεζών, των οικονομικών θεμάτων που είναι θέματα που μας απασχολούν. Δηλαδή, και από πλευράς Ευρωπαϊκής Ενώσεως και κρατών μελών θα δεχθούμε ότι είναι σοβαρή απέτηση των πολιτών και θα προβούμε σε ορισμένες επερωτήσεις προς τους πολίτες για να δούμε αν ο έλεγχος των, των χρηματοοικονομικών αγορών χρειάζεται πολιτική επέμβαση την οποία θα πρέπει να αναλάβουμε εμείς και την οποία θα μετατρέψουμε σε ένα ε, νομικό κείμενο ε, είναι θέματα για τα οποία ακόμη έχουμε αμφιβολίες και ε, πρέπει να επηρεάσουμε και την διαδικασία λήψεως αποφάσεων κατά τρόπον ώστε να ε, προωθηθεί ε, η νομική εφαρμογή αυτών των ε, πρωτοβουλειών των πολιτών. Θεωρώ ότι η πρόταση του Άντριου Νταφ είναι πάρα πολύ σωστή να καλέσουμε τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, να συζητήσουμε μαζί του και να ε, χρησιμοποιήσουμε αυτή τη δυνατότητα ε, δημοκρατικής ε, συναποφάσεως την οποία θα μοιραζόμαστε εφ' με τους πολίτες. Ζήτησε ακόμη το λόγο ο συνάδελφος Έφνερ, αλλά και εγώ θα ήθελα να σας πω τη δικιά μου γνώμη και να συμμετάσχω στη συζήτηση που ήταν πολύ ενδιαφέρουσα, ε, πολύ πλούσια. Οι παρεμβάσεις σας ανέλησαν πολύ σημαντικά θέματα που πρέπει να σημειωθούν. Και εγώ θεωρώ ότι η, ε, πρωτοβουλία των ε, πολιτών, όπως το είπε και ο κύριος Λαμασούρ αποβλέπει στο να προσεγγίσει κανείς την ε, Ευρώπη ε, προς τους πολίτες ε, και σαν Επιτροπή αναλύσαμε την απόφαση του ε, Γερμανικού Συνταγματικού Δικαστηρίου τον Ιούνιο και είχαμε πει ότι δεν αναφερόταν στην Γερμανία. Ναι, με να ε, ε, εξέταζε την Γερμανία, αλλά ουσιαστικά απασχολούσε την Ευρώπη και τον τρόπο του γίγνεσθε της Ευρώπης και γι' αυτό θέλαμε καθ' όλη την θητή αυτή να συναντηθούμε με ε, νομομαθείς ε, από όλη την Ευρώπη ξεκινώντας από τη Γερμανία διότι ε, αυτά τα θέματα άπτονται της υπάρξεως του λαού και η μεγαλύτερη επιφύλαξη η οποία υπάρχει σχετικά με την δημοκρατία στην Ευρώπη και η οποία μας καταδεικνύει ότι δεν είναι δυνατόν να καλύψουμε αυτό το δημοκρατικό έλλειμμα είναι ε, η έλλειψη ενός ε, ευρωπαϊκού λαού. Διότι ένας λαός δεν καταρτίζεται μόνο από την ιστορία αλλά και από τη συνείδηση ε, συμμετοχής σε ένα λαό και την παράδοση η οποία μεταφέρεται από τη μία γενιά στην άλλη. Οπότε η πρωτοβουλία αυτή των πολιτών θα πρέπει να μας δώσει τη δυνατότητα να αποδείξουμε ε, ότι υπάρχει ένας ευρωπαϊκός λαός. Ορισμένοι αναφέρθηκαν στο παραδεκτό. Σωστά. Αυτό το θέμα πρέπει ε, να αντιπαραταχθεί ε, στις επιπτώσεις, στα αποτελέσματα, διότι αναλόγως των επιπτώσεων που θα έχουμε σχετικά με την ε, ε, λαϊκή αυτή πρωτοβουλία, το αποτέλεσμα μπορεί να είναι πολύ σημαντικό. Και εφόσον μιλάμε για αιτήσει, άπαξε μιλάμε για αιτήσει, εξετάζουμε αν είναι ε, παραδεκτές ή όχι. Αρκεί λοιπόν να σκεφτούμε ότι εάν ε, οι αιτήσει ε, το, οι λαϊκές θα υποχρέωναν ε, την, Ευρώπη, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να απαντήσει ή προς ποια κατεύθυνση. Δηλαδή αρκούν για να ξεκινήσει μια νομοθετική διαδικασία, διότι το άρθρο 11 δεν λέει ότι το αντικείμενο της πρωτοβουλίας αυτής είναι ε, νομοθεσία. Μιλάμε για νομικά θέματα, άρα υπάρχουν ε, λεπτές έννοιες, διότι όσο πιο σαφείς θα είναι οι νομικές επιπτώσεις, τόσο μεγαλύτερος θα πρέπει να είναι και ο έλεγχος ο οποίος θα διεξάγεται. Θεωρώ ότι η έκθεση Σεύκοβιτς ε, είναι μία έκθεση η οποία είναι μεν λογική, αλλά εάν ελέγχουμε κατά τον ίμιση την ε, διαδικασία στο ίμις του χρόνου τη διαδικασία των υπογραφών ε, θα έχουμε σπαταλήσει χρόνο. Η διαδικασία αυτή πρέπει να γίνει στην αρχή και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι το όργανο που θα αποφασίσει το παραδεκτό. Η πρόταση του κυρίου Νταφ μου, λέει, ε, μου φαίνεται πολύ ενδιαφέρουσα διότι θέτει και ένα πρόβλημα όχι τόσο αρχικού ελέγχου αλλά συνεχών ελέγχων Δηλαδή, Ποιος θα πει αν έχουμε επιτύχει ε, τον σωστό αριθμό, αν επετεύχθη αυτός ελεύθερα, αν οι εθνικοί οργανισμοί θα ε, μεταβιβάσουν ε, τα πορίσματα στους, στους διεθνείς οργανισμούς. Διότι αντιλαμβάνουμε ότι η πρόταση DAF είναι μεν ενδιαφέρουσα, αλλά πρέπει να δούμε πώς θα γίνει. Διότι σε ορισμένα κράτη όπως η Ιταλία θα πρέπει να ανατίθεται ο έλεγχος σε ε, κάποιο δικαστήριο, το οποίο όμως θα επιβαρύνει κάποιο, κάποιο όργανο το οποίο ήδη έχει ευξημένες ευθύνες. Εγώ θα προτιμούσα καταρχήν να υπάρχει μία σοβαρή εξέταση που δεν θα γινόταν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά από ένα τρίτο ανεξάρτητο όργανο και πιστεύω ότι χρειάζεται οι γενικές γραμμές να διέπουν την οργάνωση και κάποιο όργανο να αναλάβει την ευθύνη, να υπερασπιστεί τη σημασία τους ε, για να αποφασίσουμε ή όχι περί του παραδεκτού. Και σε περίπτωση συζητήσεως θα πρέπει να προβλεφθεί κάποια επιτροπή, ε, διότι θα υπάρξουν ε, διάφορες ε, ε, πρωτοβουλίες που θα διατυπώνονται και θα τσακώνται μεταξύ τους πια προπορεύεται. Άρα αν υπάρχει μία επιτροπή θα μπορεί να προβεί σε ένα πιο ενδελεχή έλεγχο και θεωρώ ότι κατά αυτόν τον τρόπο θα πρέπει να τονίσουμε την ύπαρξη ενός ευρωπαϊκού λαού και θα πρέπει να στηριχθεί από τις δομές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η στήριξη αυτή πρέπει να είναι οικονομική, Αναρωτιέμαι, φοβάμαι αυτή την οικονομική ε, στήριξη γιατί φοβάμαι ότι ο και καλυμμένος στόχος θα είναι να έχουν ορισμένα ποσά στη διάθεσή τους για την επίτευξη πολιτικών στόχων και αυτό με τρομάζει. Θα έπρεπε λοιπόν να υπάρχει μια απόδειξη σοβαρότητος στις πρωτοβουλίες και για να μπορέσει ένας λαός να αναπτυχθεί χρειάζεται βοήθεια. Και σκέφτομαι την ε, βοήθεια από τα μέσα ενημέρωσης που είναι πολύ σημαντική, δηλαδή η πρωτοβουλία των πολιτών άπαξ και επιτύχει έναν ορισμένο αριθμό ε, υπογραφών θα πρέπει να γίνει γνωστή. Ε, θα πρέπει να υπάρξει ενημέρωση εγώ λοιπόν σκέφτομαι ότι πρέπει να υπάρχει και οικονομική κάλυψη και κάλυψη από πλευράς των μέσων ενημέρωσης. Γι' αυτό και θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Χέφνερ και στη συνέχεια να ρωτήσω από τον εισηγητή αν θέλει να απαντήσει. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν θα ε, αναφερθώ τώρα μόνο στις τελικές σας αλλά και στα αρχικά ερωτήματα, διότι νομίζω ότι θέσατε τον δάκτυλο του τύπου των ύλων. Δηλαδή ότι θα υπάρχει ένα μέσο να δείξουμε ότι υφίσταται ένας ευρωπαϊκός λαός και αυτή είναι μία από τις δύο ουσιαστικές διαστάσεις που, περι, ε, που περιγράφει το θέμα αυτό το οποίο συζητάμε. Δηλαδή, καταρχήν το ένα είναι ότι θέλουμε να δημιουργήσουμε έναν ευρωπαϊκό λαό αν διασύνοριακά συμμετέχουν άνθρωποι σε πολιτικές πρωτοβουλίες και τεκτενόμενα. Πράγμα που δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή και αυτό θα είναι πολύ σημαντικό διότι μέχρι στιγμή συζητάμε χωριστά στην Ελλάδα, στη Γαλλία, στη Δανία, στη Γερμανία. Δεν έχουμε μία διαευρωπαϊκή ή πανευρωπαϊκή συζήτηση για ορισμένα θέματα. Μία πρωτοβουλία λοιπόν η οποία θα διεξάγεται ε, συγχρόνως σε διάφορα μέλη της Ευρώπης μπορεί να οδηγήσει και τους λαούς να αναλάβουν κοινέ πρωτοβουλίες. Και αυτό είναι και το θέμα της δημοκρατίας. Δηλαδή οι άνθρωποι να αντιληφθούν ότι είναι η δικιά μας Ευρώπη και εγώ μπορώ να επηρεάσω. Η φωνή μου εισακούεται. Δεν υπάρχει κάποιο εκεί πάνω που κάνει ό,τι θέλει και εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Όλοι μας μπορούμε να διατυπώσουμε προτάσεις που θα εισακουστούν. Και νομίζω ότι αυτά είναι τα δύο βασικά στοιχεία. Τώρα, μεταξύ άλλων, ζήτησα το λόγο, διότι πολλές φορές η συζήτηση δεν αναφέρεται μόνο σε συγκεκριμένα θέματα, αλλά αναφέρεται και γενικότερα σε θέματα δημοκρατίας, άμεσης δημοκρατίας και από αυτού θα ήθελα να σχολιάσω ένα θέμα και να σας πω εκ προημίου ότι στη συνέχεια της συζήτησης τόσο στην Επιτροπή όσο και όταν θα υπάρξει έκθεση θα πρέπει να προσέξουμε να περιγράφουμε επακριβώς ό,τι συζητάμε και να παραμένουμε στο θέμα μας. Διότι εδώ μιλάμε γενικώ ε, για την ελεύθερη δημοκρατία, άμεση δημοκρατία, για τα δημοψηφίσματα στην Ιταλία, για την κατάσταση στην ε, Ελβετία, δηλαδή θέματα τα οποία είναι σχετικά, αλλά παραδείγματος χάρη, αν λάβουμε υπόψη τις Ηνωμένε Πολιτείε, την ε, Καλιφόρνια, όπου δεν ε, υπάρχει άμεση δημοκρατία παρά μόνο σε 22 πολιτείες. Ε, στην Καλιφόρνια όλα τα θέματα τα οποία είναι πρώτα στην επικαιρότητα είναι τα οικονομικά. Γιατί, διότι εδώ και πριν από 100 χρόνια ε, ε, καταρτίστηκε μία νομοθεσία η οποία διατύπωσε ε, μία κακή νομοθεσία στην Ελβετία. Τα λεφτά δεν είναι σημαντικά. Μπορεί η μία πλευρά να είναι πλούσια, η άλλη όχι και να κερδίσει ο φτωχός. Γιατί, γιατί οι Ελβετοί φρόντισαν άπαξ και υπήρξε ο αριθμός των υπογραφών να σταλούν τα υπέρ και τα κατά της προτάσεως σε κάθε πολίτη και ο καθένας να κρίνει μόνος του. Άρα το αποτέλεσμα είναι τελείως διαφορετικό στην Ελβετία και θα μπορούσαμε έτσι να σχολιάσουμε και άλλες χώρες. Δεν μπορούμε να αποφασίσουμε με ένα ναι ή ένα όχι. Όταν μιλάμε για νομοθεσία πρέπει να υπάρχουν έξυπνες νομοθετικές προτάσεις ε, και η δημοκρατία είναι ακριβώς ο λαός να μπορεί να συμμετέχει όρθον δυνατόν περισσότερο στην πολιτική. Θα ήθελα όμως να σας πω εδώ ότι δεν μιλάμε για λαϊκή ετοιμικορία. Δεν μιλάμε για τα, ε, ε, τις δυνατότητες που έχουν άλλες χώρες, αλλά για μια μορφή που δεν υπάρχει πουθενά μέχρι σήμερα. Δηλαδή δεν υπάρχει τίποτα που μπορεί να μοιάσει με την πρωτοβουλία των πολιτών της Ευρώπης και γι' αυτό ανησυχώ και θα σας πω ποια είναι η ανησυχία μου. Για αυτή, σε αυτή τη διαδικασία όσο πιο ισχυρή είναι αυτή η δυνατότητα πρωτοβουλία των πολιτών τόσο πιο εύκολα θα είναι κανείς να την καταχραστεί. Και θα μπορούσα να αναφερθώ ας πούμε στην Βόρειο Λινανία Βεσφαλία όπου έχουμε πολλές πρωτοβουλίες, μπορούμε να συγκεντρώσουμε υπογραφές αλλά ε, το Κοινοβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να ασχοληθεί με το θέμα ενώ στην Αυστρία μπορεί κάτι να ζητήσει κάτι και ε, είναι τελείως ελεύθερη η κυβέρνηση εάν θα το ακολουθήσει ή όχι. Χρησιμοποιούνται λοιπόν λαϊκίστικες ε, επεμβάσεις οι οποίες δεν καταλήγουν πουθενά. Ε, πιέζει κανείς μια κυβέρνηση συγκεντρώνοντας υπογραφές χωρίς όμως να καταλήξει σε τίποτα. Ενώ όπου μπορεί να ε, επιβάλλει κανείς μια απόφαση δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Χρειάζεται να υπάρχει μία αιτιολογημένη πρόταση, κάτι το οποίο δεν είναι εύκολο να γίνει, στη Γερμανία τουλάχιστον. Αυτό το οποίο φοβόμασταν όλοι, δεν έγινε ποτέ, απλώς συζητείτε. Και όταν συζητείτε, απλώς συζητάμε αν συνάδει με το Σύνταγμα ή όχι ε, αλλά εδώ μιλάμε για ένα no man's land στο ευρωπαϊκό δίκαιο το οποίο θα πρέπει να φροντίσει να είναι ναι μεν σαφές αλλά και ανοιχτό. Θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί γιατί ε, όσοι συμμετέχουν στο νομοθετικό έργο, ε, στο Κοινοβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο Συμβούλιο θα πρέπει να προχωρήσουν πολύ προσεκτικά χωρίς να ε, αναφερόμαστε σε ποια θέματα μπορεί κανείς να διατυπώσει πρωτοβουλία αλλά θα πρέπει να συνάδει με τα θεμελιώδη δικαιώματα της Ευρωπαϊκής Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπάρχουν και άλλα θέματα τα οποία θα πρέπει να συζητήσουμε λεπτομερώς. Τέλος, θα ήθελα να αναφερθώ σε δύο θέματα. Καταρχήν την ανησυχία η οποία διατυπώθηκε από τόσα σχόλια και επαναλαμβάνω και πάλι ότι η, εμπειρική, η εμπειρία μας μας δείχνει ότι όχι μόνο δεν πρέπει να φοβόμαστε τις πρωτοβουλίες των πολιτών διότι συμβάλλουν στη συμμετοχή των πολιτών η οποία είναι πολύ πιο σωστή. Είναι και ε, ένα πανεπιστήμιο πανεπιστήμιου για τους πολίτες θα έλεγα. Δηλαδή δεν πρέπει να σκεφτεί κανείς απλώς ότι υπάρχει ε, μία πολιτική από την βάση υβριστική αλλά μία συμμετοχή στη λήψη των αποφάσεων και ανάληψη ευθυνών που θα είναι προς όφελος όλων. Με συγχωρείτε, αλλά τώρα ξέχασα τι θέλω να σας πω. Υπάρχει ακόμη ένα θέμα. Ε, υπάρχει η προκατάληψη. Όταν δηλαδή ε, λένε ότι αν ψήφιζαν ε, οι πολίτες για τη φορολογία δεν θα υπήρχε φορολογία. Αλλά η εμπειρία μας έδειξε ότι όπου οι πολίτες συναποφασίζουν για τη φορολογία, διότι πολλές φορές η φορολογική νομοθεσία δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς τη συνένεση των πολιτών, ε, αποδίδει ένα σύστημα πιο διάφανο, πιο κατανοητό, πιο διάφανο, πιο κοινωνικά σωστό και ε, πιο ηθικά καλύτερο. Δηλαδή θα πληρώσουν περισσότερους φόρους εάν ε, πιστέψουν πραγματικά ότι σωστά τους ζητούνται. Ίσως λοιπόν θα έπρεπε να εξετάσουμε αυτές τις θέσεις. Δηλαδή, ε, αν η πολιτική δεν πρέπει να διατυπώνεται από κοινού με τους πολίτες για να έχουμε καλύτερη πολιτική. Ουσιαστικά όμως αυτό που θέλω να ζητήσω είναι ότι αφού ασχοληθούμε με όλα αυτά τα υψηλά θέματα, τα προβλήματα που τίθενται από τις λεπτομέρειες που απαρίθμησαν όλοι, δεν μπορούν ε, να επιληθούν βάσει ενός ερωτηματολογίου σχετικά με τα νομοθετικά όργανα τα οποία δεν υφίστανται. Διότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε καμία πρόταση ε, που να επιτρέπει τους πολίτες να αποφασίσουν για το ευρωπαϊκό γίγνεσθε, αλλά απλώς να διατυπώνουν οι πολίτες ε, πρωτοβουλίες τις οποίες ε, κατά την κρίση Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, θα γίνονται αποδεκτές ή όχι. Ευχαριστώ. Έχω ζητήσει και άλλη το λόγο. Μέσες Σμιτ πρώτα και μετά θα δώσω το λόγο στους ηγητές. Και ο κύριος Τερνέιρο ζήτησε το λόγο από την Κομισιόν. Καλά είναι, καλό είναι να μιλήσει και αυτό. Λοιπόν, πρώτο ο κύριος Μέσσερσμιτ, μετά η Κομισιόν και μετά οι εισηγητέ. Στον κύριο Νταφ ένα σχόλιο για τους περιορισμούς των πιθανών προτάσεων. Για τη θανατική ποινή. Δεν νομίζω ότι κανείς θα θέλει να αλλάξει τον κανονισμό στον τομέα αυτό. Εγώ όχι το κύριο πρόβλημα που ανακύπτει είναι αν αποκλείουμε τέτοιες προτάσεις υποτεθείς ότι αυτές οι προτάσεις δεν βγάζουν ένα εκατομμύριο υπογραφές. Αν λέμε ότι δεν μπορεί να υπάρχουν ε, οι προτάσεις που περιορίζουν υφιστάμενα δικαιώματα, μπορεί να υπάρχουν ένα εκατομμύριο πολίτες που να προτείνουν την επέκταση των δικαιωμάτων Φερρυπίν για το χάρτη. Ε, δείτε ας πούμε τι γίνεται με την ΕΣΔΑ. Συζητήσαμε το θέμα αυτό σήμερα και είπαμε ότι δεν θα, δεν θα καλύπτουν, δεν θα είναι κοινωτικό και όλα τα πρωτόκολλα. Αν πρωτο, προ, προκύψουν πρωτόκολλα στο μέλλον και δεν είμαστε σε αυτά, έχουν το δικαίωμα ένα εκατομμύριο πολίτε να δηλώσουν ότι θα πρέπει η Ένωση να προσχωρήσει και στα συγκεκριμένο πρωτόκολλο. Απ' την άλλη μεριά, Μήπως θα έχουν το δικαίωμα να πούν ότι Κάποια, που έχουμε κάποια πρωτόκολλα που έχουμε επικυρώσει δεν πρέπει να, είναι... να τα επικυρώσουμε. Δηλαδή είναι το ίδιο και το αυτό. Ε, το θετικό δικαίωμα δεν μπορεί να το δώσει αν δεν δώσει και το αρνητικό δικαίωμα. Πρέπει να έχουμε και μία εμπιστοσύνη στους πολίτες στους οποίους δίνουμε το δικαίωμα αυτό. Και μετά θα ψηφίσουμε με βάση τη συνείδησή μας. Αυτή είναι η βασική συζήτηση εδώ. Το κρίσιμο κατά την άποψή μου που πρέπει να αλλάξουμε στο κείμενο κατά απόψή μου, στην πρόταση της Επιτροπής δηλαδή, είναι το 4-4, άρθρο 4 παράγραφος 4, που αναφέρει προτάσεις που είναι προδήλως αντιφατικές προς τις αξίες της Ένωσης, πρέπει να αλλάξει και να λέμε μόνο πρωτοβουλίες που υπάγονται στις αρμοδιότητες της Ένωσης μπορούν να ε, εξεταστούν. Διότι αν αρχίσουμε να συζητάμε τι είναι αξία της Ένωσης και τι δεν είναι, θα σημαίνει ότι ορισμένε προτάσεις, κυρίως διεύρυνση δικαιωμάτων, δεν μπορούν να είναι εφαρμοστές, αλλά άλλες όχι. Άρα, δείχνουμε με τον τρόπο αυτό ότι δεν έχουμε την εμπιστοσύνη στους πολίτες αλλά όχι σε αυτούς μας που καταψηφίζουμε τις προτάσεις που, που αναφέρουν. Είναι λοιπόν σημαντικό, πολύ σημαντικό, να μην περιορίσουμε τις προτάσεις που μπορούν να προκύψουν από ένα εκατομμύριο πολιτών, να τους δείξουμε εμπιστοσύνη και να δείξουμε εμπιστοσύνη και στους εαυτούς μας. Ευχαριστώ. Ο κύριο Τρακόφσκι. Θέλω να επανέλθω σε ένα σημείο μετά τις συζητήσεις που ακούσαμε η όλη ιδέα είναι να μην απογοητεύονται οι πολίτε αν απορρίπτονται οι πρωτοβουλίε του. Ένα λοιπόν σημαντικό θέμα είναι να πούμε στο κείμενο σαφώς ότι αν κάτι δεν ανήκει σε κοινοτική αρμοδιότητα, δεν τηρεί για παράδειγμα την αρχή της επικουρικότητας, η αίτηση αυτή απορρίπτεται. Να θέσουμε σαφείς κανόνες απόρριψης και να τους διαφημίσουμε κιόλας για να το ξέρουν όλοι. Αυτό είναι πρακτικό. Ωστόσο, στη συζήτηση αυτή ερχόμαστε πίσω στο βασικό ερώτημα του ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Ποιος αποφασίζει ότι η Ένωση έχει αρμοδιότητα για κάτι. Και επανέρχομαι σε αυτό γιατί είναι προβληματικό. Έχουμε, όταν έχουμε προβλήματα με το Μάστρικτ, με την Καλσούη, όλοι πιστεύουν είναι για το, την υπεροχή του κοινοτικού δικαίου. Όχι. Είναι για το ποιο λέει, ποιο έχει αρμοδιότητα. Και αυτό το αποφύγαμε με έναν επικοδομητικό διάλογο μεταξύ του ΔΕΚ και των συνταγματικών δικαστηρίων των κρατών μελών. Αυτό όμω είναι το μείζον ζήτημα ανησυχία. Αν επανέλθουμε στο πρόβλημα αυτό, Φερρυπίν, αν αμφισβητηθεί η απόφαση τη επιτροπή, κάποιοι λένε ότι πρέπει να υπάρξει ένα ιδιαίτερο θεσμικό όργανο που θα λύνει το ζήτημα αυτό. Ποιο όργανο το ΔΕΚ που έχει μια κάποια νομιμοποίηση, α συμφωνήσουμε από αυτού, έχει προβλήματα. Πάντα έναντι των συνταγματικών δικαστηρίων. Αν εμφανιστεί και άλλο όργανο, θα έχει ακόμα μικρότερη νομιμοποίηση. Αυτό λοιπόν πρέπει να το πούμε σαφώ. Να το διαφημίσουμε. Βέβαια μετά υπάρχει το ερώτημα τι γίνεται αν μια τέτοια αίτηση προχωρήσει. Τι κάνουμε αυτή. Δεύτερη ερώτηση. Απαιτεί αλλαγή των συνθήκων. Τι κάνουμε. Να το σκεφτούμε αυτό. Λέει η Κομισιόν, ε, τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να υποβάλουμε μια πρωτοβουλία που απαιτεί αλλαγή συνθήκη. Να ζητήσει αυτό το Συμβούλιο να προχωρήσει και να λάβει θέση. Το ίδιο και η επικουρικότητα. Έχουμε εμπιστοσύνη ότι η Επιτροπή μπορεί να το αποφασίσει αυτό. Εγώ έχω. Αλλά Το καταλαβαίνει ο κόσμος. Να λέμε ότι αυτό είναι επικουρικότητα, άρα ε, δεν τίθεται. Αυτή είναι η άποψή μου. Πρώτα να το διαφημίσουμε, να το δημοσιοποιήσουμε και δεύτερον να ε, ξέρουμε ακριβώς ποια είναι αυτά τα θέματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Ωραιότατα. Δίνω το λόγο λοιπόν στον εκπρόσωπο της Επιτροπής τώρα. Oui, merci, Monsieur le Président. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Οι εισηγητά, κύριε και κύριε εισηγητές. Πολύ ενδιαφέρουσε οι παρατηρήσει όλων των μελών. Θέλω, δεν θα τι σχολιάσω, απλά να διευκρινίσω κάποια σημεία που θεωρώ σημαντικά για την συνέχεια των συζητήσεων. Το θέμα του ελέγχου από τα κράτη-μέλη. Το σύστημα που προτείνει η πρόταση δεν ξεκινά από ιδεολογικά απριόρι, αλλά από, ρεαλιστική, από μια ρεαλιστική προσέγγιση. Εάν θέλουμε να έχουμε ένα νομοθετικό κείμενο για την άσκηση των δικαιωμάτων αυτών γρήγορα, θεωρούμε ότι ο έλεγχος των υπογραφών μπορεί να γίνει μόνο από τα κράτη-μέλη. Γι' αυτό, ε, για ρεαλιστικούς λόγους προτείνουμε αυτή τη θέση. Δεν μπορούμε να το δούμε αγίως. Για τους ελέγχους παραδεκτού. Πριν ε, φτάσει στην Επιτροπή. Να διευκρινίσω κάποια πράγματα. Δεν υπάρχει μόνο έλεγχο του παραδεκτού μετά τι 300.000 υπογραφέ μόνο. Δημιουργείται ένα ολόκληρο σύστημα που βοηθά τους διοργανωτέ τη πρόταση και φιλτράει τρόπον την, την πρωτοβουλία αυτή. Πρώτον, καταχωρείται η πρωτοβουλία αυτή πριν ξεκινήσει η, η, η συλλογή υπογραφών, καταχωρείται στην Επιτροπή που Τη δίνει με τον τρόπο αυτό και κάποια έτσι υποστήριξη επιμελητιακή, δηλαδή ε, ενημέρωση ας πούμε. Η Επιτροπή στη φάση αυτή ήδη θα έχει αν χρειαστεί ένα διάλογο με τον οργανωτή για να διευκρινίσει σημεία που είναι σαφή. Τη στιγμή της καταχώρησης λοιπόν, αν ο στόχος της πρωτοβουλίας είναι σαφής, η Επιτροπή θα προσπαθήσει να το διευκρινίσει με, τον, ε, υπεύθυνο, τους υπεύθυνους πριν προχωρήσει παραπέρα. Αυτό είναι σημαντικό. Τελευταίο σημείο. Υπάρχουν δύο κατηγορίες φίλτρων ταυτόχρονα πριν την καταχώρηση. Η Επιτροπή μπορεί να μην καταχωρήσει αν η πρόταση είναι παράλογη ή προδήλωσα βάσιμη και κάτι πολύ σημαντικό επίσης, αν η πρόταση είναι αντίθετη με τις αξίες Ένωσης. Αυτό αφορά παραδείγματο χάρη πρωτοβουλίες ε, επαναφοράς της θανατικής ποινή. Ήδη εξ αρχής δηλαδή η πρωτοβουλία αυτή ούτε καν θα καταχωρείται. Θα απορρίπτεται διότι για παράδειγμα η θανατική ποινή θεωρείται ότι είναι αντίθετη μεταξύ της Ένωσης. Όταν μιλάμε για παραδεκτό το επίπεδο των 300.000 υπογραφών, για ένα θέμα και μόνο μιλάμε που δεν είναι εύκολο. Το κατά πόσον υπάρχει στη συνθήκη νομική βάση ή όχι για να προτείνει η Επιτροπή αυτό που τη ζητείται να προταθεί. Η πρόταση της Επιτροπής είναι να βρει μια ισορροπία Πολλοί είχαν ζητήσει η ανάλυση αυτή να γίνει στο ξεκίνημα. Άλλοι ωστόσο είχαν πει ότι δεν πρέπει να αρχίσει τη λογοκρισία από νωρί η Επιτροπή. Από την άλλη υπάρχει κίνδυνος να πνιγεί η Κομισιόν από χιλιάδες ε, αιτήσει. Αν απαιτείται για κάθε αίτηση να γίνεται έτσι εμπεριστατωμένη νομική ανάλυση. Απ' την άλλη πλευρά δεν μπορούμε να περιμένουμε μέχρι το τέλος για να μην ε, αυξήσουμε τις προσδοκίες των πολιτών και για να μην υποχρεώσουμε τα κράτη-μέλη να αρχίσουν να κάνουν ελέγχους των υπογραφών για κάτι που εν τέλει θα κρίνει η Επιτροπή επίσημα ότι ήταν απαράδεκτο. Προφανώς η πρόταση είναι συζητήσιμη, αλλά η φιλοσοφία, είχε, η φιλοσοφία της ήταν να υπάρξει μια εξισορρόπηση μεταξύ μιας πολύ πρώιμης και πολύ καθυστερημένης ανάλυσης. Αυτή ήταν η φιλοσοφία της Επιτροπής. Ό,τι αφορά το όργανο, η, αν το όργανο προσφυγής, ας πούμε, η απόφαση της Επιτροπής ε, εξετάζεται προφανώς από την δυνατότητα των διοργανωτών της πρωτοβουλίας να προσφύγουν στο ΔΕΚ. Μπορεί να υπάρχουν, να, να, να, θέλουμε άλλα προβλήματα, αλλά προφανώς ε, είναι αρμοδιότητα του ΔΕΚ, γιατί πρόκειται για μια απόφαση που βλάπτει, που θίγει τους διοργανωτές. Και το δικαστήριο είναι το μόνο όργανο που εν τέλει μπορεί να, να κρίνει, γιατί πρόκειται περί de facto συνταγματικού ε, δικαστηρίου αν το, η απόφαση είναι νομότυπη ή όχι. Αυτά. Ευχαριστώ. Λοιπόν, οι συγγητές θέλουν το λόγο. Το λόγο, κύριος Λαμασούρ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε. Ευχαριστώ για την πολύ καλή ποιότητα της συζήτησης και την ε, εξαιρετικά ε, ενδιαφέρουσα σειρά παρατηρήσεων που ακούσαμε. Θα είμαι σύντομος. Συμφωνώ μαζί σας κύριε Πρόεδρε και με τους περισσότερους συναδέλφους ότι ο έλεγχος παραδεκτού πρέπει να γίνεται αμέσως. Αυτή η ιστορία των 300.000 υπογραφών, κατά την άποψή μου, δεν πιστεύω ότι θα λειτουργήσει. Είναι πανάκριβο, γραφειοκρατικό και δεν στέκει. Πρέπει, όταν θέλει κάποιο να ξεκινήσει μια πρωτοβουλία, να γνωρίζει εξ αρχή κατά πόσο είναι παραδεκτή ή όχι βεβαίως υπό τον έλεγχο του, του ΔΕΚ με προσφυγές. Όπως προτείνεται πρέπει να υπάρχει κάποιο δικαιοδοτικό όργανο που γνωμοδοτεί, διαφορετικό κατά την από την Κομισιόν, ο καθένας έχει το ρόλο του. Κάτι που πρέπει να εφεύρουμε. Εγώ προσωπικά ωστόσο είμαι πολύ επιφυλακτικός ε, σε σχέση με το σύστημα που προτείνει η Κομισιόν. Συμφωνώ με τη γενική φιλοσοφία της πρότασης, με πολλές από τις τεχνικές λεπτομέρειες, αλλά δεν νομίζω ότι στέκει έτσι όπως είναι. Επίσης, συμφωνώ με την πρόταση DAF να ακούσουμε την άποψη του διαμεσολαβητή μας, του κ. Διαμαντούρου, που την ξέρει την κατάσταση και άλλωστε συνεργάζεται στενά και η Επιτροπή Αναφορών μαζί του. Ας ρωτήσουμε λοιπόν κατά πόσον μπορεί να παίξει ένα ρόλο είτε στην επίσημη διαδικασία είτε στην παράλληλη διαδικασία που περιέγραψα νωρίτερα. Να στέλνουμε δηλαδή στο διαμεσολαβητή όσου δεν πληρούν α, ε, τους όρους της χρήσης της βασιλικής οδού. αλλά που θα ήθελαν να έχουν και μια πιο συγκεκριμένη απάντηση στα αιτήματά τους. Επίσης είναι χρήσιμο, όπως αναφέρθηκε από τον συνάδελφο κύριο Γκερέρο να υπάρξει διαβεβαίωση για την, για την οικονομική διαφάνεια όσων ξεκινούν την πρωτοβουλία. Αν είναι λόμπι πρέπει να το ξέρουμε. Αν δεν είναι λόμπι πρέπει να ξέρουμε πώς χρηματοδοτούνται. Υπάρχει χρηματοδότηση της πρωτοβουλία. Υπάρχει κατόπιν η χρηματοδότηση συλλογή υπογραφών που προφανώ είναι αρμοδιότητα ε, των κρατών μελών. Είναι σαφές ωστόσο ότι πρέπει να γνωρίζουμε ποιος κρύβεται πίσω από την ΑΒ πρωτοβουλία. Κάτι σημαντικό για μένα είναι ότι ο κύριος στόχος της νέας αυτής πρωτοβουλίας δεν είναι να δώσουμε σε πολιτικά κόμματα που δεν μπόρεσαν να πετύχουν το στόχο τους, είτε εδώ είτε σε εθνικό επίπεδο, να με άλλο μέσο να πετύχουν το, το στόχο τους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να περάσουν μέσω της πρωτοβουλία. Βεβαίως μπορεί να χρησιμεύσει σε κάτι τέτοιο. Όπως στην Επιτροπή Αναφορών βλέπουμε ότι ορισμένε συλλογικέ αναφορές ήταν ε, ψευδό αναφορές. Στην πράξη ήταν αναφορές, ήταν παρεμβάσει ενός πολιτικού κόμματος. Προφανώς θα συμβεί κάτι τέτοιο. Αλλά δεν είναι αυτός ο στόχος της πρωτοβουλίας δεν είναι ένα επιπλέον όργανο εργαλείο των πολιτικών κομμάτων και όπως έλεγε ο κύριος Γκέρο θα πρέπει να είναι όχι ένα μέσο για να υπάρξει ανταγωνισμός της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας αλλά συμπλήρωμα και να ακουστούν οι πολίτες αυτός είναι ο στόχος που δεν ακούει κανείς διότι δεν έχουν εδαφικά την, κριτική, την κρίσιμη μάζα που θα τους επέτρεπε να ακουστούν από τους πολίτες, γιατί βρίσκονται σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να σα δώσω κάποια παραδείγματα. Στο οικογενειακό δίκαιο. Ποιο ενδιαφέρεται για τα διεθνικά ζευγάρια που έχουν το ένα παιδί τους που γεννήθηκε στην τρίτη χώρα, μένουν στην τέταρτη χώρα και που κάποτε πεθαίνει ο ένας, συγχωρίζουν και δημιουργούν απίθανα προβλήματα ε, επιτροπίας, κληρονομικά κλπ. Ποιο ενδιαφέρεται για αυτά τα θέματα. Ευτυχώ υπάρχει σήμερα μία επίτροπο, η κυρία Ρέντινγκ, που ανέλαβε το ζήτημα που άρπαξε τον τάβρο από τα κέρατα. Να σα δώσω ένα παράδειγμα. Η Γαλλία δεν αναγνωρίζει τον γάμο των ομοφυλόφιλων. Η λογική συνέπεια, η λογική νομική συνέπεια αυτού είναι ότι ένας Γάλλος που συνάπτει ένα γάμο με έναν ομόφυλό του εκτός Γαλλίας. Στη Γαλλία ο γάμος του δεν αναγνωρίζεται, γιατί εκεί δεν υπάρχει τέτοιος γάμος. Λογικό αυτό. Αυτό που είναι τελείως παράλογο και σκανδαλώδες, θα έλεγα ότι αν δύο Βέλγοι, δύο Ολλανδοί, δύο Ισπανοί του ιδίου φίλου παντρεύονται νόμιμα στη χώρα τους, δεν αναγνωρίζεται παρά αυτά και αυτόν όνο γάμος στη Γαλλία. Δεν αναγνωρίζει δηλαδή η Γαλλία την κυριαρχία του Βελγίου στο θέμα του οικογενειακού δικαίου έναντι Βέλγων πολιτών. Αυτό είναι ασύλληπτο. Θέτουμε λοιπόν στους ανθρώπους ε, περιορισμούς που είναι άσχετους. Άλλο θέμα. Οι υπότροφοι Εράσμους που διαπιστώνουν ότι όταν πάνε σε δύο-τρία πανεπιστήμια της Ευρώπης διαφορετικά σε διαφορετικά χώρες, τα διπλώματά τους δεν αναγνωρίζονται στη χώρα όπου παίρνουν το δείπνο. Αυτό είναι απαράδεκτο, αντιβαίνει στο γράμμα κοινοτική νομοθεσίας, αλλά είναι το 0,7% των, ε, του εκλογικού σώματο εμά. Οπότε ποιο νοιάζεται για τους φοιτητέ Εράσμους. Άλλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι ίδιοι συνολικοί διακινούμενοι. Φορολογικά, εργατικά, αστικά, οικογενειακά προβλήματα κλπ. Τα ζητήματα αυτά δεν τα λαμβάνουν υπόψη τα πολιτικά κόμματα. Η διαδικασία αυτή λοιπόν έχει ως πρώτο κύριο στόχο, όχι μοναδικό, να δώσει στους πολίτες εκείνους στους οποίους κανείς δεν ενδιαφέρεται, να ακούσουν το δικαίωμα να ακουστούν. Μπορεί να είναι πάνω από ένα εκατομμύριο στην Ένωση. Αλλά κανείς δεν ενδιαφέρεται για τα δικαιώματά τους. Για τα θέματα τώρα. Ανεξάρτητα από τα θέματα που ενδιαφέρουν τους πολίτες, υπάρχουν και πολιτικά θέματα που θα τεθούν. Είτε για να παρέμβει η Ένωση σε ένα τομέα, είτε για να σταματήσει να παρεμβαίνει ή να αλλάξει την παρέμβασή της. Είναι προφανές και το λέει η συνθήκη ότι παραδεκτές θα είναι μόνο οι πρωτοβουλίε που ανήκουν σε, σε ενωσιακή αρμοδιότητα. Αυτό που είπε και ο κύριος Σμιτ, για να μην μπαίνουμε στο θέμα των αξιών της Ένωσης επί μακρόν, πλην όμως, προσοχή, ο χάρτης των θεμελιωδών δικαιωμάτων προφανώς απαγορεύει τη θανατική ποινή στην Ένωση και σε όσες χώρες έχουν υπογράψει την ΕΣΔΑ, αλλά το δικαίωμα στη ζωή που είναι στο άρθρο 1 του χάρτη, σε κάποιες χώρες σημαίνει ότι ερμηνεύεται ως απαγορευτικό της άμβλωσης, ενώ σε άλλες χώρες ως επιτρέπον την άμβλωση. Το ίδιο ισχύει και με πολλές άλλες αξίες. Άρα το μόνο στέρεο νομικό αγκυροβόλιο για μας είναι οι αρμοδιότητες της Ένωσης. Από εκεί και πέρα όμως θα αντιμετωπίσουμε προτάσεις, πιθανές προτάσεις, ενδεχομένως που μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα. Ο κ. Γκερέρο μίλησε για τα δημοσιονομικά θέματα. Εγώ δεν είμαι τόσο αισιόδοξο ο κύριο Χέφνερ που λέει ότι όποτε ζητάμε από τον κόσμο να ψηφίσει φόρους, ο, ο κόσμος τους ψηφίζει. Δείτε τι γίνεται στην Καλιφόρνια από την πρόταση, δεν ξέρω τι νούμερο που ψηφίστηκε στην Καλιφόρνια, η Καλιφόρνια έχει φαλυρίσει μόνιμα. Δεν υπάρχουν φόρες στην Καλιφόρνια πια. Σκεφτείτε, σκεφτείτε, τέτοια εποχή που είμαστε, να υπάρξει ένα εκατομμύριο πολιτών που ανήκουν σε χώρες που συμβάλλουν στον κοινοτικό προπολογισμό να ζητήσουν μείωση του κοινοτικού προπολογισμού. Επίφοβο ζήτημα, αυτό είναι αρμοδιότητα της Ένωσης μπορεί να πείτε ότι δεν είναι αρμοδιότητα τη Ένωση. Ομοίω. διεύρυνση. Τι γίνεται εκεί. Η διεύρυνση της η διεύρυνση τη Ένωση δεν είναι αρμοδιότητα τη Ένωση, είναι επέκταση τη Ένωση μέσω διεθνού συνθήκη. Αλλά από τη στιγμή που λέμε ξεκινάμε τι ενταξιακέ διαδικασίε με μία χώρα, την Κροατία, α πούμε, την Κροατία, συγγνώμη, α πούμε, και υπάρχουν κάποιοι πολίτες που δεν τη θέλουν την Κροατία. Θα μπορούσαν κάλλιστα να αντιταχθούν, να αντιταχθούν, συγγνώμη, στο ξεκίνημα των, ε, στην έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων. Βλέπετε τι πολιτικά προβλήματα μπορεί να τεθούν. Η συνθήκη δεν προβλέπει η πρωτοβουλία αναφορά αφορά τροποποίηση τη συνθήκη. Με μια μεγάλη συζήτηση που είχαμε με την έκθεση Κάουφμαν και που ανέφερε ο κ. Νταφ προηγουμένω. Βεβαίω! Αλλά για την κατανομή των ευρών μεταξύ χωρών τη Ένωση. Αυτό είναι παράγωγο δίκαιο. Αρμοδιότητα τη Ένωση. Σκεφτείτε. Ένα εκατομμύριο πολιτών να λένε εγώ δεν μπορώ να ζήσω σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση όπου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν υπάρχει αναλογική εκπροσώπηση των πολιτών. Ή διαφωνώ με την αρχή της φθήνουσας αναλογικότητας που περιλαμβάνει η συνθήκη. Και το τι θα πει φθήνουσα μπορούμε να το ερμηνεύσουμε όπως θέλουμε. Αυτό είναι, αυτό σημαίνει να μπαίνουμε σε ένα θεσμικό ζήτημα. Δεν είναι να ασχολούμαστε με ένα συγκεκριμένο κεφάλαιο μιας συνταξιακής διαδικασίας. Τελευταίο παράδειγμα, γιατί σας είπα ότι θα είμαι σύντομος. Τι γίνεται αν έχουμε μπροστά μας δύο ή περισσότερες αντιφατικές πρωτοβουλίες για, τις, ε, για τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς. Από τη μια μεριά έχει κάποιου που θέλουν να κάνουν πιο σκληρή την κοινωτική νομοθεσία για αυτό το ζήτημα και έχει άλλο ένα που λένε σταμάτα να μα ζαλίζετε πια με του ε, γενετικά τροποποιημένου οργανισμού. Τι θα κάνουμε. Τι σημαίνει αυτό. Μήπως με τη σημερινή συζήτηση θα έπρεπε εμείς ή η Κομισιόν, κάποιος, ένα όργανο που δεν θα είναι η Κομισιόν, αυτός ο δικαιοδοτικός ε, το όργανο της πρώτης προσφυγής πριν την δεύτερη προσφυγή στο ΔΕΚ, θα έπρεπε να δώσει ή να φτιάξει έναν καθοδηγητήριο, ε, τέλος έναν οδηγό, έναν κώδικο, τα παραδείγματα που αναφέρω δείχνουν τη δυσκολία του προβλήματος. Γιατί σε κάθε ζήτημα υπάρχει η νομική διάσταση και η πολιτική κρίση. Δεν διευκολύνει το πρόβλημα έτσι, αλλά δείχνει ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη τα διάφορα αυτά στοιχεία και τις διάφορες πιθανότητες για να είμαστε βέβαιοι ότι προσφέρουμε απαντήσεις σωστά από την αρχή που είναι η πιο ενδεδειγμένη για να απαντήσει. Άρα μήπως έπρεπε να κάνουμε έναν κώδικα. του παραδεκτού. Αυτές είναι οι πρώτες γρήγορες παρατηρήσεις μου σε πρώτη φάση, πρόεδρε. Η συζήτηση δείχνει πόσο ενδιαφέρον είναι το θέμα και πόσο περίπλοκο αν θέλουμε να έχουμε ένα σύστημα αποτελεσματικό. Ευχαριστώ. Πήρατε τις παρατηρήσεις μας, δείξατε πόσο σύνθετο είναι το ζήτημα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε στους γιατί πρέπει να υλοποιήσουμε τη συνθήκη της Λισαβόνας. Και άλλο συζήτηση θα γίνει και εσείς θα δουλέψετε περισσότερο. Η κυρία Γκουρμάη. Λοιπόν, ας διευκρινίσουμε για όλους μας ότι η συνθήκη για μας στο Κοινοβούλιο πρέπει να καταρθίσει το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα λειτουργήσει αυτή η πρωτοβουλία. Θα πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε ότι υπάρχουν δύο ουσιαστικά αρχές ε, στην πρόταση αυτή. Καταρχήν ότι πρέπει να υπάρχει αντιπροσωπευτικότητα των συμφερόντων της ενώσεως, πράγμα το οποίο είπαν πολλοί συνάδελφοι είναι της αρμοδιότητας μας και ότι θα είναι εύκολο στη χρήση ε, και στον χρήστη, πράγμα το οποίο δεν είναι προφανές. Θα ήθελα λοιπόν να σας πω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε πολύ σωστή δουλειά. Ε, όχι μόνο διότι έκαναν πάρα πολλές διαβουλεύσεις όπως είπε ο κύριος Έφνερ, οργάνωσαν την ε, δημόσια ακρόαση και κατά τη συζήτηση αυτή διατύπωσαν μία σαφή πρόταση η οποία είναι ε, ήδη μία πρόταση των ε, πολιτών μας. Ας σκεφτούμε λοιπόν πόσοι πολίτες έχουν διαβάσει τις συνθήκες γιατί αν διαβάσετε τη συνθήκη θα ξέρετε τι είδους πρωτοβουλίες μπορείτε να αναλάβετε. Πρέπει λοιπόν εμείς να δώσουμε κάποια κατεύθυνση ως προς τη διατύπωση του πλαισίου. Ο πολίτης θα πρέπει να καταλάβει ότι έχει τη δυνατότητα τώρα να καλύψει αυτό το δημοκρατικό έλλειμμα, να το μειώσει και θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ σαφείς και να έχουμε μία πολύ απλή διατύπωση. Βέβαια είναι μια ευκαιρία την οποία όμως θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε συνολικά και γι' αυτό με τα μεγάλης χαράς διαπίστωσα ότι πολλοί συνάδελφοι έχουν επίσης κάνει σχόλια ε, για να σας πω ότι τώρα πρέπει να υπάρξει και μία τρίτη δυνατότητα ιστορική για τους Ευρωπαίους πολίτες και να εξασφαλίσουμε ότι θα είναι προς όφελος των πολιτών, διότι όλο και λιγότεροι ε, ψηφοφόροι πολίτες Ευρωπαίοι συμμετέχουν στις ευρωεκλογές. Οπότε θα πρέπει ε, σαν εκπρόσωποι της Ευρώπης να προσπαθήσουμε να αναβιώσουμε αυτή την Ευρώπη και θα πρέπει να είμαστε πολύ σαφείς ως προς την Ευρώπη την οποία προσφέρουμε. Έχουμε μια καλή νομοθεσία, έχουμε ε, διάφορους ε, έμπειρους οι οποίοι διατυπώνουν αυτήν την νομοθεσία για να βελτιώσουμε τη λειτουργία της Ευρώπης που θα πρέπει να διευκρινιστεί επίσης και πέραν αυτού θα πρέπει να υπάρχει μία σαφής παραδοχή και να ξέρουμε πώς θα προχωρήσουμε στη συνέχεια. Να είμαστε σαφείς σε αυτά που θα πούμε ή τους πολίτες. Συμφωνώ ότι χρειαζόμαστε ορισμένες υπογραφές για να ε, μπορέσουμε να ε, διαπιστώσουμε ε, αν η πρόταση λειτουργεί σωστά ή όχι και είναι ε, κάτι που πρέπει να γίνει στην αρχή κατά τρόπον ώστε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να θα κάνει τη δουλειά διότι αν έχουμε εκατοντάδες χιλιάδες προτάσεις και δούμε ότι δεν θα λειτουργήσουν αντιλαμβάνουμε ότι ο λόγος για τον οποίο θέλετε να έχετε 300.000 ε, ε, υπογραφές εγώ ελπίζω ότι θα χρειαστούν λιγότερες Γι' αυτό είπε ο φίλος μου επικεφαλής της Επιτροπής Προϋπολογισμού ότι πρέπει να το δούμε και από πλευράς προϋπολογισμού. Ε, δεν είναι θέμα το ένα εκατομμύριο των υπογραφών, αλλά είναι ότι οι υπογραφές αυτές θα πρέπει να εξυπηρετήσουν την Ευρώπη και να βαίνουν προς τη συστή κατεύθυνση, να μην εξυπηρετούν πολιτικά συμφέροντα, αλλά να βελτιώνουν την Ευρώπη για όλους, για τους ε, ε, αναπήρους για ε, όλους και θα πρέπει να το συζητήσουμε με τους συναδέλφους θα έχουμε και τον Πάολο από τη Γραμματεία για να μας καθοδηγήσει και να δούμε πώς θα διατυπώσουμε την καλύτερη δυνατή πρόταση. Και εσείς αγαπητοί συνάδελφοι έχετε τη δυνατότητα να μας βοηθήσετε. Και χαίρομαι που είναι εδώ η ε, Προεδρία, εκπροσωπείται εδώ η Προεδρία διότι στην ε, Τρόικα έχουν συζητήσει πολύ για αυτό το θέμα και θα πρέπει να καθορίσουμε και το χρονοδιάγραμμα για την ε, ομάδα που θα το αναλάβει αλλά θα πρέπει να παραμείνουμε συνεπείς για να βελτιώσουμε την Ευρώπη προς όφελος όλων μας. Ευχαριστώ. Είναι 18 και 30. Άρα ε, κλείσαμε τη συζήτησή μας και αύριο θα συναντηθούμε σε 9 το πρωί. Καλό βράδυ.